good morning. Um, Καλημέρα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την, να ξεκινήσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Κάποιοι από εσά μπορέσατε να παρακολουθήσετε χθε μία παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό IUU. Κάποιοι που μπόρεσαν να είναι παρόντες εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερως. Περίμενα την Κομισιό να μας πει πόσο καλά δουλεύει ο κανονισμός και πόσο πίεση ασκείται από τη, στη μία και στην άλλη χώρα να αλλάξουν τις πρακτικές τους, πόσο πίεση ασκείται να υιοθετήσουν σωστές πρακτικές με βάση τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών. Τα έχουμε ακούσει αυτά και στο παρελθόν. Και μετά περίμενα να δοθεί ο λόγος στι μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίες θα έλεγαν ότι δεν κάνουμε αρκετά και ότι όλα αυτά είναι ωραία λόγια και τίποτα άλλο. Το αντίθετο συνέβη. Οι ΜΚΟ είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει εξαιρετική δουλειά και σημειώνεται πολύ σημαντική πρόοδος, κάτι το οποίο μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Να βλέπουμε δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή τη δυνατότητα να επιφέρει αυτή τη συνεργασία έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση με την ε, λαθρέα λία. Παράνομη και το καθεξής. Σήμερα το πρωί έχουμε τον κύριο Κομ Λόρντεν από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας το οποίο, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το συμβούλιο, το ISIS, Συνεχώ μιλούμε για το ISIS, το Διεθνέ Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της ε, Θάλασσας, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο τα και γιατί τα επιστημονικά δεδομένα ποικίλουν από τη μία χρονιά στην άλλη, με συνέπειες ενίοτε αρκετά δύσκολες ε, για τους ενδιαφερομένους. Σας δίνω ευθύ αμέσω το λόγο, κύριε Κόλμ Λόρντεν. Κύριε Αντιπρόεδρε του Διεθνούς ε, Συμβουλίου αυτού, θα έχετε PowerPoint από ό,τι φαίνεται και θα μας κάνετε την παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, παρουσίαση αυτή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα που παρουσιάζω το ΆΙΣΙ στο Διεθνές Συμβούλιο σήμερα σε εσάς, την Επιτροπή σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω <laughs> No, not working. Ευχαριστώ. Να σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες για τον εαυτό μου, για να ξέρετε και ποιος μας μιλάει. Εγώ είμαι επιστήμονες στον τομέα της αλίας, από, από πάντα θα έλεγα ήμουν ένθερμος ο υπέρμαχος της θάλασσας από έφηβος ε, ασχολούμαι με αυτά τα θύματα, με απασχολεί Φορεία. και για το κατά πόσο ξέρουμε αν τα αποθέματα είναι βιώσιμα ή όχι. Με ενδιαφέραν πάντοτε τα θέματα της βιολογίας, των ηχθειοαποθεμάτων. Έκανα σχετικές σπουδές που ολοκληρώθηκαν με διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Κόρκ στην Ιρλανδία και έχω 20 χρόνια εμπειρία στο Ιρλανδικό ε, ε, Ινστιτούτο για τη Θάλασσα. Έχω ασχοληθεί με τον τόνο, με την καραβίδα, με την αλία στην ανοιχτή θάλασσα, μεγάλου βάθους και στα βίνθοπερλαγικά είδη με έχω ασχοληθεί ιδιαίτερως για τα αποθέματα της Καραβίδας στη θάλασσα της Ιρλανδίας και έχω συμμετάσχει στο Διεθνές Συμβούλιο για πάρα πολλά χρόνια. Έχω συμμετάσχει σε πάνω από 70 ομάδες εμπειρογνωμών και έχω προεδρεύσει σε πάνω από 16 από αυτές τις ομάδες εμπειρογνωμών. και από τον Ιανουάριο του 2018 είμαι αντιπρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή του ΆΙΣΙΣ, στην ΑΚΟΜ και θα σας εξηγήσω αργότερα περί τίνος πρόκειται. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να σας μιλήσω για, γύρω από αυτά τα θέματα που βλέπετε στην οθόνη. Γύρω από, θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις σε αυτές τις βασικές ερωτήσεις. Τι είναι το ISIS, το Διεθνές Συμβούλιο, σε ποιο πλαίσιο παρέχει τη συμβουλευτική του υπηρεσία και θα σας μιλήσω και για τη διαδρομή ε, που ακολουθούμε για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμβουλευτική υπηρεσία. Θα σας μιλήσω για τα δεδομένα, για το πώς αξιολογούμε τα ηχθή αποθέματα, πώς ε, καταλήγουμε σε σημεία αναφοράς για τα διάφορα ηχθή αποθέματα και θα σας μιλήσω για την προσέγγιση του οικοσυστήματος στο μέλλον. Σε σχέση λοιπόν με τα σημεία αναφοράς με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, το ISIS, που ε, καταλήγει σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε επιστημονικά πορίσματα για την αηφόρο χρήση θαλασσών και ωκεανών. Είμαστε ένα δίκτυο 5.000 ειδικών και πυρογνωμόνων από 700 ιδρύματα ερευνητικά και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Και κυρίως μας ενδιαφέρει το επιστημονικό μας πεδίο, εστιάζεται κυρίως στο ε, ε βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό. 1.500 ειδικοί και εμπειρογνώμονες συμμετέχουν στις ε, συνεδριάσεις μας ετησίως. λειτουργούμε με βάση το στρατηγικό μας σχέδιο, το οποίο εκπονήσαμε και ανακοινώσαμε τον περασμένο Ιανουάριο. Θέλουμε να είμαστε μια οργάνωση η οποία να είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την επιστήμη της θάλασσας προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας για αμερόληπτη συμβουλευτική για την κατάσταση και την αηφόρο χρήση θαλασσών και ωκεανών. Θέλουμε να ε, προωθούμε την επιστημονική κατανόηση των θαλασσίων οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν. Θέλουμε να ε, χρησιμοποιούμε και να αξιοποιούμε αυτές τις γνώσεις για να καταλήγουμε σε ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου για, σε σχέση με την διαχείριση και την επίτευξη των στόχων αηφορίας. Είμαστε μία από τις πιο παλαιές διακυβερνητικές οργανώσεις στον κόσμο από το 1908 λειτουργεί το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας. Βλέπετε τις χώρες μέλη μας. Με πορτοκαλί βλέπετε τις χώρες που συμμετέχουν. Είναι η πλειονότητα της Βόρειας Ευρώπης, συμμετέχει η Ρωσία οι και η Βόρειος Αμερική, ο Καναδάς. Όλα αυτά είναι, όλες αυτές οι χώρες είναι μέλη του Διεθνού Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας και έχουμε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με άλλες χώρες και άλλες οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, στην Αρκτική, στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στη Βόρεια Θάλασσα μεταξύ άλλων. Πώς λειτουργούμε λοιπόν. Έχουμε ένα δίκτυο 5.000 εμπειρογνωμόνων, ειδικών και αξιοποιούμε τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις για να εμπλουτίσουμε το επιστημονικό πεδίο και για να μοιραστούμε και να διαδώσουμε ε, αυτή τη γνώση. Προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα στοιχεία που μας παρέχουν οι επιστήμονες έτσι ώστε να ε, χτίσουμε πάνω σε αυτά τις συμβουλές μας και θέλουμε αυτά τα στοιχεία να ανταποκρίνονται στις, στις αρχές της διαφάνειας, της δίκαιης παρουσίασης ε, της δυνατότητας να είναι αξιοποιήσιμα αυτά τα στοιχεία από όλους και προσβάσιμα από όλους. Μας ενδιαφέρει να αναπτύσσουμε εργαλεία και τεχνικές για να αναλύουμε και να αποθηκεύουμε δεδομένα. Και θα δείτε εντός ολίγου ότι έχουμε ένα ενεργό κέντρο δεδομένων μέσα στο Διεθνές Συμβουλίο για την Εξερεύνηση της, της Θάλασσας. Το ISIS ασχολείται με συνέδρια επίσης, με εργαστήρια, με κατάρτιση, με εκπαίδευση. Η οργάνωσή μας ε, πάνω σε δύο πυλώνες, τη συμβουλευτική από τη μία και την επιστήμη από την άλλη. Παράγουμε δηλαδή επιστημονικό έργο και ε, κάνουμε έρευνα πάνω στην οποία θα ε, στηριχθεί η, δραστη, η συμβουλευτική μας δραστηριότητα. Έχουμε 150 ομάδες εμπειρογνωμόνων που ε, λειτουργούν σε αιτήσια βάση, στις οποίες συνεισφέρουν με εμπειρογνώμονες και ειδικοί από πάνω από 60 χώρες. Με βάση λοιπόν το στρατηγικό μας σχέδιο, ασχολούμαστε με τα οικοσυστήματα. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε έρευνα η οποία θα εμπλουτίσει τις γνώσεις και την κατανόησή μας για το οικοσύστημα. Προσπαθούμε να αναλύσουμε τον αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στο εκάστοτε οικοσύστημα. Ε, χρησιμοποιούμε τις νέες ε, τεχνικές της παρατήρησης και της εξερεύνησης ή μάλλον για να κάνουμε παρατήρηση και εξερεύνηση χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνικές που μας προσφέρει η τεχνολογία. Αξιοποιούμε δηλαδή τις νέες, τις νέες τεχνολογίες για να διερευνήσουμε τις αλλαγές που διαπιστώνονται στον ωκεανό σε βάθος χρόνου. Ασχολούμαστε με την παραγωγή, ε, με την έρευνα σε σχέση με κάνουμε επιστημονικό έργο και ερευνητικό για την ε, παραγωγή ε, θαλασσινών. Προσπαθούμε να παρακολουθούμε δηλαδή επιστημονικά το πώς γίνονται όλες αυτές οι ηχθειοκαλλιέργειες. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε με την διαχείριση με την έρευνα σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, μας ενδιαφέρει η σχέση της θάλασσας με την ε, κοινωνία, με την ανθρώπινη κοινωνία. Πάντοτε βασιζόμαστε στις νέες τεχνολογίες. Το ISIS λοιπόν είναι ένας πάροχος γνώσης, παρέχει τη βέλτιστη δυνατή επιστημονική γνώση ως συμβουλευτική υπηρεσία σε διεθνείς και εθνικές αρχές. Παρέχουμε συμβουλές για πάνω από 240 ήχθη αποθέματα κάθε χρόνο. Παρέχουμε συμβουλές για τα παράπλευρα αλλιεύματα, για τον αντίκτυπο στα, ε, στον ωκεανό, στην ανοιχτή θάλασσα, για τα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα και βιοτόπους, για τις ε, προστατευόμενες περιοχές και ε, τα σχετικά οικοσυστήματα. Βλέπετε κάποιους φορείς τους οποίους παρέχουμε ε, συμβουλές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ε, ΟΣΠΑΡ, την ε, Επιτροπή Αλίας του Βορείου Ατλαντικού, την ΑΦΚΟ, την το ΦΑΟ, την ΑΣΚΟ, την ΑΜΚΟ και διάφορους άλλους σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς. στους οποίους παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παρέχουμε δηλαδή τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις τις οποίες πρέπει να βασιστούν οι θύνοντες για να λάβουν τις αποφάσεις, τις αποφάσεις τους. Το ISIS, όπως σας είπα, έχει ένα πολύ ενεργό και δραστήριο κέντρο δεδομένων. Συντονίζουμε όλα τα δεδομένα σε σχέση με τα θέματα και το θαλάσσιο περιβάλλον στο Βόρειο Ατλαντικό ενημερώνουμε συνεχώς το κέντρο δεδομένων μας, ε, ασχολούμαστε συνέχεια με την εμβάθυνση της επιστημονικής μας γνώσης και τρίτο σκέλος είναι ο τρόπος με τον οποίο παρέχουμε συμβουλές για την αϊφόρο διαχείριση των ηχθιαποθεμάτων. Και αυτό είναι αυτό που σας ενδιαφέρει άλλωστε. Παρέχουμε λοιπόν συμβουλές για τις ε, δυνατότητες αλλιεύματος για πάνω από 240 αποθέματα το χρόνο, για τον αντίκτυπο στα οικοσυστήματα και ε, παρέχουμε μια γενικότερη επισκόπηση και λεπτομερή ανάλυση της αλλιευτικής κατάστασης και των οικοσυστημάτων στις διάφορες περιοχές ή περιφέρειες. Ε, δεχόμαστε 30 ειδικά αιτήματα περίπου κάθε χρόνο από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, τη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον, από κάποια χώρα που μπορεί να είναι μέλος ε, του ISIS, αλλά και από άλλους ε, δικαιούχους τροποντινά, εντολοδόχους. Ασχολούμαστε δηλαδή με αιτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον αντίκτυπο της αλλιευτικής δραστηριότητας, την πίεση και τον αντίκτυπο στον πυθμένα της θάλασσας λόγω της αλλιευτικής δραστηριότητας, αιτήματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης αλλιευτικής δραστηριότητας, την αξιολόγηση των ευπαθών ε, βιοτόπων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων ή το αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στα ήχθη αποθέματα. Τα αλλιεύματα είναι ένας δημόσιος πόρος που είναι περιορισμένος, κινητός και δημόσιος. Ε, χρειάζεται λοιπόν διαχείριση. Η υπερβολική ε, εκμετάλλευση αυτού του δημόσιου πόρου οδηγεί σε μειωμένη παραγωγικότητα και ενδυνάμει, μη ενδυνάμει ζημιά που δεν δύναται να αντιστραφεί. Επίσης, η αλληλεία σε ένα κράτος μέλος έχει αντίκτυπο στις αλληλευτικές δυνατότητες σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, χρειάζεται σωστή διαχείριση. Η αλληλευτική πόρη είναι ένας δημόσιος πόρος και αυτό, ε, γι' αυτό αποκαλείται κοινή αλληλευτική πολιτική, γιατί είναι ένας κοινό πόρος που ανήκει σε όλους. Επιτρέπουμε λοιπόν στην, στον αλληλευτικό κλάδο να εκμεταλλευτεί αυτό τον δημόσιο πόρο. Άρα κάθε συμβουλευτική που δίδεται πρέπει να γίνεται αντικείμενο διεθνούς συντονισμού και διεθνούς σωστής διαχείρισης προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα αυτού του διεθνούς πόρου. Θα θέλω τώρα να περάσω στο περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε. Όλες αυτές δίδονται, δίδονται με βάση διεθνείς συμφωνίες, τις οποίες θα σας δείξω στην επόμενη διαφάνεια, και σχετίζονται και με την πολιτική των αποδεκτών, των παραληπτών, αυτών που ζητούν τη δική μας συμβουλή. Οι διάφορες επιτροπές, οι διάφορες επίσημες ε, κρατικές αρχές και το καθεξής. Στόχος μας είναι να υιοθετούμε την ε, προσέγγιση της προφύλαξης. Ε, προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε υπόψη μας τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και θέλουμε να έχουμε μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά ε, των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε. Έχουμε ε, ως βασικές συμφωνίες την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, όπου εδρεώνεται για πρώτη φορά αυτή η αρχή της βέλτιστης αηφόρου βιώσιμης απόδυσης. Έχουμε το UNCD, την διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1992, που θεσμοθέτησε την αρχή της προφύλαξης και την προσέγγιση αυτή. Έχουμε την UNFCA, τη συμφωνία λοιπόν για αυτά τα ηχθειοποθέματα του 1995 που πάλι εδραίωσε την αρχή της προφύλαξης στη Σύμβαση για τη Βιοπικιλότητα των ΗΠΑ του 1992 που υιοθέτησε την προσέγγιση του προστασίας του οικοσυστήματος και τη διακήρυξη του Johannesburg στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Εφόρο Ανάπτυξη το 2002 η οποία επικύρωσε την προσέγγιση του οικοσυστήματος και την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ε, Βεβαίω, λαμβάνουμε υπόψη μα την εθνική και περιφερειακή νομοθεσία, όπω είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι το στρατηγικό πλαίσιο, το MSFD, το, ο νορβηγικό νόμο για του θαλάσσιου πόρου, ο ομοσπονδιακό νόμο τη Ρωσική Ομοσπονδία για την Αλία, ο νόμο διαχείριση αλληλευτικών αποθεμάτων τη Ισλανδία, αλλά και ο, η αντίστοιχη νομοθεσία τη νήσου Φαρόε, μεταξύ άλλων. Πώς καταλήγουμε στις ε, ε, συμβουλές που παρέχουμε. Έχουμε την ακόμα την Συμβουλευτική Επιτροπή στο ΆΙΣΟΣ, η οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή αυτών των συμβουλών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή ανταποκρίνεται στα, αιτήματα, στα τα σχετικά αιτήματα από τις χώρες μέλη, από διεθνείς επιτροπής, από οργανώσεις, από διάφορους φορείς διαχείρισης οικοσυστημάτων και ηχθειοαποθεμάτων. αποθεμάτων. Οι συμβουλέ που παρέχουμε βασίζονται στην αρχή τη προφύλαξης και στην προσέγγιση του οικοσυστήματος, σύμφωνα με τους στόχους, του διαχειριστικού αυτών των αρχών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή δουλεύει με διάφορου ενδιαφερόμενου φορεί για να διασφαλίσει ότι οι συμβουλέ αυτέ είναι κατανοητέ και σημαντικέ για την ε, κοινωνία. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ένα πρόεδρο, τον κύριο Κικόλα, τέσσερι αντιπροέδρου, είμαι ο ένα από αυτού, και είκοσι μέλη, ένα εκπρόσωπο από κάθε χώρα μέλος. Εν συνεχεία, έχουμε και διάφορες επιτροπές και αν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ε, συζητούν για συγκεκριμένη χώρα ή αν κάποιος ας πούμε έχει συγκεκριμένες γνώσεις έρχονται ε, στη συνεδρίαση για να εγκρίνουν την ε, Συμβουλή. Οι συμβουλές Καταρχάς, η πρώτη φάση τη διαδικασία είναι ότι διατυπώνεται ένα αίτημα, η οποία ε, αναπτύσσεται στα πλαίσια επαναλαμβανόμενων διαλόγων με αυτούς που υποβάλλουν την ερώτηση και τους επιστήμονες και θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ε, ερώτηση. Συνθέτουμε την γνώση, γίνεται μια τέτοια διαδικασία, γίνεται διασφάλιση της ποιότητας, ε, χτίζουμε τη γνώση, ε, μέσω διαδικασία με συνεδριάσει εμπειρογνωμόνων και έχουμε και μια πολιτική για τα δεδομένα την οποία προσυπογράφουμε. Γίνεται μια ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης ομοτήμων, είναι σημαντικό σε επιστημονικό πεδίο. Έχουμε ανεξάρτητους ερευνητές ε, που εξετάζουν τι κάνουμε και θέλουμε να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση της ε, υπάρχουσας, των επαρχουσών επιστημονικών υπαρχόντων συγγνώμη, ε, επιστημονικών δεδομένων για τα διάφορα αποθέματα. Τέλος, παράγουμε την, τη συμβουλή, ε, συντάζουμε απαντήσεις στο ερώτημα και δημοσιεύουμε τα στοιχεία αυτά στην ιστοσελίδα μας, εξηγούμε το αιτιολογικό στη συμβουλή αυτή και οι συμβουλές αυτές γίνεται με διεθνή συνένεση στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Εδώ με περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε τα διάφορα βήματα της διαδικασίας αυτής. Έχουμε τη διατύπωση του αιτήματο. Έχουμε δύο διαφορετικά είδη συμβουλών, τις τακτικές συμβουλές για τα διάφορα ήχθη αποθέματα. Δίνουμε συμβουλές, ας πούμε, ετησίως ή μία φορά στα δύο χρόνια για αυτά τα ήχθη αποθέματα ή μπορεί να έχουμε ειδικά αιτήματα και όταν ε, υποβληθούν και συμφωνήσουμε για, αυτές τις, ε, για αυτά τα αιτήματα, πάνε στις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Αν είναι τακτικό το αίτημα αυτό, πηγαίνει σε ειδικό εργαστήρι, το οποίο συγκαλείται για να ασχοληθεί με αυτό το ειδικό αίτημα και συνεχεία έχουμε την κοινότητα των 1.500 ε, εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται με μας. Έχουμε την διαδικασία διασφάλισης ποιότητας και έχουμε ανεξάρτητες επισκοπήσεις μέσω ελέγχων που γίνονται αν είναι τακτική η συμβουλή αυτή, η παρεχόμενη συμβουλή, ή αν είναι ειδική η συμβουλή, πληρώνουμε για να γίνει ανεξάρτητη εξέταση της συμβουλής αυτής και έχουμε τη διαδικασία σύνταξης της συμβουλής, όπου μια υποομάδα της Συμβουλευτικής Επιτροπής ε, συντάσσει την τελική συμβουλή, η οποία επικυρώνεται από την ACOM, ε, την Συμβουλευτική Επιτροπή. Τώρα, η βάση της δουλειάς που κάνουμε στο ISIS είναι η συλλογή των δεδομένων. Ήθελα να το αναφέρω εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, στο σημερινό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας ε, προβλέπονται 520 εκατομμύρια ευρώ για τη συλλογή δεδομένων που ταξοδεύουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συλλέγουν όλα τα δεδομένα τα οποία πηγαίνουν στις αξιολογίες του ISIS για τις υπηρεσίες της αλίας, ε, προγράμματα δειγματοληψία στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δουλειά του ISIS, να έχουμε καλά δεδομένα, ούτως ώστε να μπορούμε να παρέχουμε συμβουλές για τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. Τα είδη των δεδομένων που συλλέγουμε θα εστιάσω καταρχάς ε, στην αξιολόγηση των ε, ηχθιαποθεμάτων, πώς την κάνουμε αυτήν την αξιολόγηση και θα σας δώσω μια γεύση για το πώς γίνεται η δουλειά μας. Ε, κάνουμε, παίρνουμε δείγματα στα λιμάνια, ε, πάνω στα σκάφη, για το μήκος, το βάρος, την ηλικία και άλλες βιολογικές παραμέτρους που είναι η οριμότητα και το φύλλο και έχουμε έτσι μια ιδέα για την το μέγεθος, τη, δημογραφική κατανομή του πληθυσμού και τις αλλαγές που συμβαίνουν συν το χρόνο και που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στην παραγωγικότητα και το περιβάλλον. Επίσης, έχουμε μια ανεξάρτητη ενημέρωση για την αλία από επιστημονικές έρευνες που είναι έρευνες στις στράτες σε διαφορετικά μέρη. Επίσης, από διάφορες μελέτες που κάνουμε στον πυθμένα της θάλασσας, χρησιμοποιούμε επίσης ακουστικές μεθόδους για να μετρήσουμε το μέγεθος του πληθυσμού των, θαλάσ... Ε, ψαριών στα μέσα της θάλασσας, επίσης και για, τις, για τα αυγά και τον για να ξέρουμε πού είναι ε, το ο αναπαραγωγικός πληθυσμός και σε τι κατάσταση που είναι, ε, σε τι κατάσταση είναι και σε τι κατάσταση είναι η βιομάζα ανάλογα με, το... με την ποσότητα των αυγών. Χρησιμοποιούμε επίσης υποθαλάσσια τηλεοπτική επισκόπηση των αποθεμάτων ε, για να δούμε ας πούμε, την κατάσταση το... της καραβίδας ας πούμε, στον πυθμένα και εκεί καταλαβαίνουμε, παίρνω μια ιδέα για την κατάσταση του πληθυσμού. Οι έρευνες γίνονται σε ερευνητικά σκάφη ε, στα διάφορα κράτη-μέλη του ISIS, αλλά συνεργαζόμαστε και με τον αλληλευτικό κλάδο για να κάνουμε αυτές τις έρευνες. Βασικό στοιχείο στην αξιολόγηση των αποθεμάτων είναι οι πληροφορίες που έχουμε από τα αποθέματα ε, τις έχουμε από το ημερολόγιο του σκάφους, από τα λιμάνια, από τα ταξίδια που κάνουν παρατηρητές, από τους κανονισμούς ελέγχου και παίρνουμε καλές πληροφορίες για το, το ποσό ψαριών που αλλιεύθηκε, για τον ε, τόπο που βρίσκονται αυτά τα αποθέματα, το, τη χρονική στιγμή και τα παραλιεύματα. Ειδικά σε, μικτές, σε μεικτά ηχθιαποθέματα, σε μεικτά αλλιεύματα. Τώρα πώς τα συνδυάζουμε όλα αυτά και καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση είναι το απόθεμα. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε απευθείας τον, και με ακρίβεια τον πληθυσμό. Έμεσα τον να υπολογίζουμε με βάση τα δεδομένα ε, για, το βόρειο για τη Βόρεια Θάλασσα, ας πούμε. Κάνουμε έμεσους υπολογισμούς του μεγέθους του χθιαποθέματος. Κοιτάμε καταρχάς το, τη ε, δομή, το μέγεθος του πληθυσμού, πόσα είναι τα... Στην αρχή έχουμε πολλά μικρά ψάρια, καθώς ε, μεγαλώνουν, κάποια πεθαίνουν φυσικά και όσο γυράσκουν μειώνονται ακόμα περισσότερο και έχουμε πολύ λιγότερα μεγάλα ψάρια το παρακολουθούμε αυτό σύντο χρόνο και βλέπουμε τις αλλαγέ στο μέγεθος και στη δομή του πληθυσμού και αυτό μας δείχνει το ποσοστό θνησιμότητας του αποθέματος και τις αλλαγέ στην ανανέωση του πληθυσμού, που είναι ο αριθμό δηλαδή των γόνων που μπαίνουν και ανανεώνεται ο πληθυσμό. Ο βαθμός θνησιμότητας, όπως είπα, είναι η αλλαγή στον αριθμό ε, λόγω της ηλικίας και η θνησιμότητα προκαλείται είτε από φυσικούς παράγοντες είτε από την αλληλεία. Ο πληθυσμός πεθαίνει, υπάρχουν παράσιτα. Φυσικά χρειαζόμαστε να έχουμε καλές μετρήσεις για τα αλλιεύματα, ούτω ώστε να ξέρουμε ποια είναι η βιομάζα του ηχθιαποθέματος, το μέγεθος του πληθυσμού σε κάθε φάση. Αν έχουμε ένα πληθυσμό μας στον ωκεανό, κάποια μικρά, κάποια μεγάλα ψάρια ας πούμε, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο απόθεμα το οποίο προσωπείται εδώ από το πράσινο ε, δίχτυ ε, που αφαιρεί ας πούμε ένα τμήμα του πληθυσμού σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό κάθε χρόνο. Έχουμε τις πληροφορίες από το μυρολόγιο του σκάφους που μας δίνει πληροφορίες για το μέγεθος των αλλιευμάτων. Έχουμε δειγματοληψία ε, στα αλλιεύματα αυτά που πιάνουμε και βλέπουμε συνολικά τι εκφορτώνεται από τον ε, πληθυσμό του ηχθιαποθέματος και έχουμε και έρευνες που μας δείχνουν που μας δείχνουν ανεξάρτη, ανεξάρτητο τρόπο ε, τον τρόπο που ανανεώνεται ο πληθυσμός και συνδυάζουμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να παράγουμε μοντέλα αξιολόγησης του αποθέματος, όπως τα λέμε, που είναι μαθηματική εκπροσώπηση του τι συμβαίνει στη φύση. Και αυτές οι εκτιμήσεις προσπαθούν να μας δώσουν μία πραγματική εικόνα για το μέγεθος του πληθυσμού και τη σχέση ανάμεσα ε, στο απόθεμα και στο μέγεθος του πληθυσμού ε, για να μάθουμε το... τη θνησιμότητα. Γίνονται διάφορες αξιολογήσεις του αποθέματος ε, στον ΆΙΣΙΣ ανάλογα με τις πληροφορίες που έχουμε και την καταλληλότητα των μοντέλων αυτών αξιολόγησης των ηχθιαποθεμάτων. Ε, να ξεκινήσω με τα δεδομένα, από εκεί που ξεκίνησα. Όλα αυτά βασίζονται σε καλά δεδομένα. Εάν τα δεδομένα δεν είναι επαρκή, δεν είναι συνεπή μεταξύ του ακριβή, οποιοδήποτε μοντέλο, α πούμε, δεν, δεν αξίζει, θα προσπαθήσει να μας δώσει την εικόνα του πληθυσμού, του αποθέματος, αλλά από σαθρά δεδομένα. Όταν μιλάω για δεδομένα, ο κόσμος δεν ε, καταλαβαίνει με τι μοιάζουν αυτά τα δεδομένα. Προσπαθώ να σας δείξω εδώ με τι μοιάζουν τα δεδομένα. Αριστερά βλέπουμε την κατανομή των ε, εκφορτώσεων από τις έρευνες, ε, από την... Από Ισλανδικά ψάρια, το μπακαλιάρο της Ισλανδίας, από το 95 ξεκινήσαμε, μέχρι το 19 έχουμε στοιχεία. Ο Εγγελφίνος πιο συγκεκριμένα. Ε, βλέπετε κάποια ανώτατα όρια ας πούμε, στον πληθυσμό συν το χρόνο. Για κάποιους λόγους, μέσα σε αυτά τα χρόνια, βελτιώθηκαν τα κατάσταση των αποθεμάτων και δεξιά βλέπετε γραφικές παραστάσεις ε, με βάση τη χρονική ηλικία, όχι με βάση το μήκο. Βλέπουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλα σμήνη ψαριών. Βλέπουμε αδύναμα επίσης σμήνη σε κάποιες φάσεις. Όταν έχουμε καλά στοιχεία στα δεδομένα, έχουμε πολύ σαφή εικόνα για την αξιολόγηση, όπως παραδείγματος χάρη για την αγγελφίνο της Ισλανδίας. Άρα λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των αξιολογήσεων των αποθεμάτων που κάνουμε. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη ρέγγα της Βορείου Θάλασσας. Έχουμε λοιπόν εδώ τα αλλιεύματα ε, για τα οποία υπάρχουν διάφορε διακυμάνσει, δηλαδή στα τέλη της δεκαετία του 1970 είχαμε μια μεγάλη μείωση ε, των αλλιευμάτων ε, και γύρω στο μισό εκατομμύριο τόνους τώρα ε, είναι ο μέσος όρος των αλλιευμάτων. Μετά στα δεξιά βλέπουμε ε, την μέτρηση σε ό,τι αφορά το recruitment, δηλαδή τα νέα μικρά σε ηλικία ψάρια τα οποία προστίθενται στον υφιστάμενο πληθυσμό και βλέπετε τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά τη Ρέγκα στη Βόρειο Θάλασσα. Βλέπουμε και τη συσχέτιση δηλαδή που υπήρξε δηλαδή. Ακριβώς επειδή υπήρξαν, υπήρξε μικρός αριθμός των νέων νυχθείων τα οποία προσθέθηκαν στα υφιστάμενα ε, αποθέματα είχαμε αυτή τη μεγάλη μείωση στην αλληλεία στα τέλη της δεκαετίας του 70 ενώ τώρα βλέπουμε να έχει υπάρξει ανάκαμψη αλλά στα τελευταία χρόνια και πάλι η προσέλευση των νέων νυχθείων έχει μειωθεί και πάλι. Τώρα κάτω αριστερά βλέπουμε ε, τη μέτρηση της ε, αλευτικής δηλαδή το ποσοστό των των πληθυσμών ή, εν πάση περιπτώσει, ένα, το τμήμα εκείνο το, το, των νυχθείων το οποίο ε, εξάγεται από τον εφισταμένο πληθυσμό. Και βλέπετε δηλαδή εδώ και την ε, σύγκριση με το επίπεδο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, ε, δηλαδή το τι ακριβώς προβλέπουμε ως ελάχιστο όριο για το ΣΕΦΠΕ. Πρόεδρος, μπορώ να σας διακόψω για ένα λεπτό και να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή μας λέτε ότι, και το βλέπουμε και στο, στο, στο διάγραμμα εδώ, ότι στα τέλη της δεκαετίας του 70 ακριβώς δεν υπήρξε χαμηλή προσέλευση νέων ηχθείων στο απόθεμα, μειώθηκε πολύ η αλληλεία. Ποια είναι λοιπόν η συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεγέθη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, είναι απάντηση, που επηρεάζουν την, ε, την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, εάν έχουμε ε, μείωση ακριβώς της, της προσθήκης των νέων εκτίων θα πρέπει να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να ανακάμψει αυτή η προσθήκη των νέων εκτίων ε, στο, στο υφιστάμενο απόθεμα και θα σας δείξω σε λίγο τι ακριβώς εννοούμε αλλά σε ό,τι αφορά διάφορα αποθέματα ε, ότι όταν έχουμε, βρισκόμαστε κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο σε ό,τι αφορά τον όγκο του αποθέματο, αυτό σημαίνει ότι ακριβώ έχουμε χαμηλή προσέλευση νέων νυχθείων και κατά συνέπεια θα πρέπει να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να ε, διασφαλίσουμε τη διατήρηση του αποθέματο. Ο πρόεδρο λέει, άρα λοιπόν η αναπαραγωγή ε, είναι όταν μα λέτε η προσθήκη αυτών των νέων νυχθείων, έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα λοιπόν η αλληλεία επηρεάζει αυτή την αναπαραγωγή. Όχι αυτό μπορεί να οφείλεται και στην αλία ή και στο όχι. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μπορεί να υπάρχει υπεραλίευση, δηλαδή αλλιεύουμε περισσότερο από όσο μπορεί να αναπαράγεται και να αντικαθίσταται ε, το, ε, το απόθεμα. Δηλαδή, εάν υπεραλλιεύουμε για σειρά ετών, τότε ε, μειώνεται λογικά το απόθεμα, αλλά υπάρχουν και περίοδοι διακοιμάνσεις, δηλαδή φυσικές σε ό,τι αφορά την ε, αναπαραγωγή, δηλαδή την προσθήκη νέων ηχθείων, σε ορισμένε περιόδου είναι χαμηλότερη, σε άλλε περιόδου είναι υψηλότερη. Οπότε σε περιόδου ακριβώ όπου έχουμε χαμηλότερη ε, προσθήκη νέων νυχθείων, θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα για να διατηρούμε το απόθεμα στα βιώσιμα επίπεδα. Αλλά εάν μου επιτρέψετε. Εμ... Θα σα δείξω στι επόμενε διαφάνειε το τι ακριβώ μπορούμε να κάνουμε. Ναι, λέει ο πρόεδρο, να μα εξηγήσετε πώ μπορούμε να πιέσουμε τα ε, ψάρια να αναπαραχθούν περισσότερο. Απάντηση. Ε, όχι, αυτό που μπορούμε να επηρεάσουμε εμεί από την πλευρά μα είναι η θνησιμότητα, δηλαδή η αλεύση. Δεν μπορούμε δηλαδή να ε, επηρεάσουμε κατά κάποιο τρόπο την ε, δυναμική εξέλιξη ε, τη αναπαραγωγή του. και δεν μπορούμε για παράδειγμα να επηρεάσουμε και την φυσική θνησιμότητα των ηχθείων. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για διαχείριση των αποθεμάτων, μιλάμε για διαχείριση τη αλληλεθνική θνησιμότητας, δηλαδή τη θνησιμότητας των ηχθείων λόγω τη αλληλεία και τίποτα παραπάνω. Ωραία, συνεχίζω λοιπόν. Τώρα σε ό,τι αφορά τα προληπτικά ε, μέτρα, ε, σημεία αναφορά. Ε, δηλαδή, σε σχέση ακριβώ με το ερώτημα που θέσατε, θα πρέπει να διατηρούνται τα εφιστάμενα αποθέματα εντό ασφαλών βιολογικών ορίων. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν παρεμποδίζεται η επιτυχής αναπαραγωγή. Βλέπετε δηλαδή ότι εάν έχουμε μικρότερο απόθεμα, έχουμε και μικρότερη προσθήκη νέων νυχθείων. Όταν έχουμε μεγαλύτερο απόθεμα, περισσότερου νέου νυχθεί οι οποίοι προστίθεται. Οπότε εξετάζουμε και τον όγκο, το, το μέγεθο δηλαδή, και ε, την ε, ε, προσθήκη των νέων νυχθείων για να δούμε ποια είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου αποθέματο. Και θέλουμε δηλαδή να διασφαλίζουμε ακριβώ αυτό, ότι δεν υπάρχει εμπόδιο σε ό,τι αφορά την επιτυχή αναπαραγωγή, δηλαδή την προσθήκη νέων νυχθείων, στο απόθεμα. Και Ε, επειδή ακριβώ αυτό το διαπιστώνουμε με βάση την, ε, την, την παρατήρηση των αποθεμάτων σε βάθο χρόνου, πάντω δίνουμε και ένα περιθώριο ε, για να είμαστε σίγουροι ακριβώ ότι δεν βρισκόμαστε κάτω από αυτό το όριο. Τώρα, για παράδειγμα, εδώ σα δίνω ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά το ε, γάδο ε, τη ε, Βορείου Βλέπετε δηλαδή εδώ στα αριστερά το ελάχιστο όριο και στα δεξιά βλέπετε μία πράσινη γραμμή σε αυτό το διάγραμμα που ξεκινάει δηλαδή από το σημείο αναφοράς και, και πηγαίνει προς τα δεξιά. Δηλαδή, από εκεί και μετά έχουμε τις ε, ε, υψηλότερη ε, την νυχτή, την υψηλότερη αναπαραγωγή δηλαδή σε αυτό το απόθεμα ε, του γάδου. Ενώ στα δεξιά βλέπουμε την κόκκινη γραμμή όπου υπάρχει αυτό το υψηλότερο σε κίνδυνος να μην υπάρχει δυνατότητα ε, διατήρησης του αποθέματος. Άρα λοιπόν εκεί στα δεξιά έχουμε ακριβώς το οριακό σημείο αναφοράς το οποίο δηλαδή ε, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αναπαραγωγική ικανότητα του, του αποθέματο. Και προσπαθούμε ακριβώ λοιπόν ποτέ να μην υπάρχει, να μην πηγαίνουμε κάτω από αυτό το μπιλίμα, αυτό το όριο δηλαδή αναφορά. Από εκεί και μετά υπάρχει και ένα άλλο όριο αναφορά, το οποίο είναι το BPA, δηλαδή η βιομάζα που βρίσκεται πάνω από το κατώτατο όριο που είπαμε το B-LIM. και όπως είπατε και εσείς στην αρχή οι αξιολογήσεις σε ό,τι αφορά τα αποθέματα των νυχθείων είναι εκφύσεως αβέβαιες. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα αρκετά υψηλότερο περιθώριο πάνω από το οποίο θα βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το BLIM. Με 95 δηλαδή τις 100 ε, ε αυτό το BPA μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν, σε καμία περίπτωση ακόμα και με την αβεβαιότητα στις αξιολογήσεις δεν βρισκόμαστε κάτω από το BLIM σε κάθε δηλαδή περίπτωση θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα περιθώρια να διατηρούμε ε, την, ε, τα αποθέματα πάνω από το πύλιμ σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο λαμβάνουμε υπόψη μας είναι το ότι θέλουμε να έχουμε την μέγιστη δυνατή απόδοση από, τους, από τα διάφορα αποθέματα. Δηλαδή, το, έχουμε μια σειρά από διατροφικά στοιχεία και πρωτεΐνη που αντλούμε από τους εχθείς, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να αλλιεύουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε αυτή την τροφή στο, τα τρόφιμα στους πληθυσμούς μας. Οπότε υπάρχει ε, μια θεωρητική καμπύλη σε ό,τι αφορά την ε, απόδοση της ε, αλληλείας. Δηλαδή, όπως, όσο ανεβαίνει η αλλιευτική θνησιμότητα, αρχίζει αυτή η καμπύλη να αυξάνεται, αλλά καθώς αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο η αλληλευτική προσπάθεια, φτάνουμε στην επωνομαζόμενη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Αν υπερβούμε αυτό το σημείο της μέγιστης βιώσιμη απόδοσης, το απόθεμα ε, αρχίζει να μειώνεται, να μειώνεται όλο ένα και περισσότερο μέχρι που να καταρρεύσει εντελώ. Άρα λοιπόν η μέγιστη ε, βιώσιμη απόδοση είναι ακριβώς αυτός ο στόχος, δηλαδή να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αναπαραγωγική ικανότητα του εν λόγω αποθέματος. Τώρα μπορούμε να εξετάσουμε το ίδιο σύστημα από μια άλλη οπτική γωνία. Στα δεξιά λοιπόν βλέπετε πάρα πολλά αλλιευτικά σκάφη αλλά πολύ μικρό μέγεθος αποθεμάτων και πολύ ε, χαμηλά λεύματα Αυτή είναι η κατάσταση δηλαδή στην οποία μπορούμε να βρεθούμε μέσω τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, δηλαδή όπου αρχίζει να φτάνει κοντά στο σημείο κατάρρευση, δηλαδή εξαφάνιση του συγκεκριμένο απόθεμα. Και σιγά σιγά περνάμε τώρα προ τα αριστερά, όπου βλέπουμε στην ε, δεύτερη εικόνα δηλαδή από τα δεξιά ε, ε, μάλλον στη δεύτερη από τα αριστερά, λιγό, πολύ λιγότερα αλλιευτικά σκάφη, πολύ ψηλότερο απόθεμα και πολύ περισσότερα αλλιεύματα και αυτό είναι ο στόχος μας όταν ε, εκπονούμε τα διάφορα ε, ε σχέδια διαχείρισης της αλληλείας. Και στο πρώτο εικονίδιο βλέπουμε πάρα πολύ λίγα αλλιευτικά σκάφη, πάρα πολλά αποθέματα και λίγα λιεύματα, πράγμα το οποίο είναι καλό για το περιβάλλον, αλλά δεν είναι καλό σε ό,τι αφορά την λευτική παραγωγή. Πρόεδρο, μπορώ να σας διακόψω και πάλι. Ναι, γιατί αναφερόμαστε συνέχεια στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αυτό το MSY. Ναι, βλέπουμε αυτή την ε, διαφάνεια, δηλαδή αν έχουμε μόνο ένα ε, αλλιευτικό σκάφο και έχουμε πολλά αποθέματα, όταν έχουμε περισσότερα αλλιευτικά σκάφη, τότε ε, μπορούμε να έχουμε περισσότερα αλλιεύματα και μπορούμε, μας λέτε, να το κάνουμε βιώσιμα. Αλλά γιατί δεν, δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα αλλιευτικά σκάφη. Ε, όπως, ε, δηλαδή, σε αυτή, την πρώτη, σε, αυτό, σε αυτή την πρώτη εικόνα της διαφάνειας. Ε, και να έχουμε, δηλαδή, ταυτόχρονα πολύ υψηλά αποθέματα και αλλιεύματα. Απάντηση. Γιατί όσο περισσότερα αλλιευτικά σκάφη έχουμε, τόσο μικρότερα γίνονται τα αποθέματα και τα αλλιεύματα. Εντάξει, δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε σε αυτό, δηλαδή ως προς το πώς μπορείτε ακριβώς να διαχειριστείτε την αξιοποίηση των φυσικών σας πόρων. Δηλαδή θέλετε να έχετε μόνο ένα αλλιευτικό σκάφος ε, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη ε, αλλιευτική ικανότητα ή θέλετε να έχετε περισσότερα αλλιευτικά σκάφη με χαμηλότερη ε, αλλιευτική ικανότητα το καθένα. Αυτό είναι δηλαδή μια ένα τεχνικό αν θέλετε ζήτημα ε, πολιτικής και όχι καθαρά επιστημονικό ζήτημα. Ε, εξαρτάται δηλαδή και από το ποιο έχει και ποια ποσόστοση και ούτω καθεξής. Ε, σε ό,τι αφορά πάντως την ε, προσέγγιση του οικοσυστήματος θα πρέπει να κάνουμε το εξή. Ναι, μεν η μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι καλή, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε ε, στην περίπτωση όπου αυτή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση οδηγεί για παράδειγμα σε ε, ζημίες ε, σε ό,τι αφορά τον ε, πυθμένα ή για παράδειγμα έχει καταστροφικές συνέπειες σε ό,τι αφορά τα ε, πτηνά, ε, τα παράκτια πτηνά και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτή την προσέγγιση των οικοσυστημάτων. Τι κάνουμε λοιπόν για να παράσχουμε συμβουλέ σε ό,τι αφορά τα αλλιεύματα του επόμενου έτου. Με βάση λοιπόν τι αξιολογήσει των αποθεμάτων που κάνουμε και την ε, ιστορική εξέταση τη εξέλιξη των αποθεμάτων, γιατί είδατε στι προηγούμενε διαφάνειε ότι εξετάζουμε ιστορικά ακριβώ τη θνησιμότητα, την αλλιευτική, ε, την αναπαραγωγική ε, και το, την βιομάζα του αποθέματο αναπαραγωγή. Βλέπουμε πώ θα διαμορφωθούν, για παράδειγμα, στο 2020 τα εν λόγω αποθέματα. Γιατί ακριβώ σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή στην εκπόνηση των συμβουλών για τα αποθέματα του 2020. Άρα λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας την οριμότητα, ε, το ποσοστό ανάπτυξης, ε, τον, ε, την, την προσθήκη νέων νυχθειών, την, τις επιπτώσεις των αλλιευτικών εργαλείων, τους φυσικούς θανάτους και ό,τι καθεξής και μετά κάνουμε μία σειρά από υπολογισμό σενάριων ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί από, πρόθεσμα το απόθεμα και από εκεί και μετά κάνουμε και υπολογισμού σε ό,τι αφορά την μέσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εξέλιξη των αποθεμάτων, για να δούμε δηλαδή πώ θα εξελιχθούν στο μέλλον τα αποθέματα. Τώρα, πώ το ISIS παρέχει αυτές τις συμβουλές. Υπάρχει καταρχήν μια ιεραρχία. Έχουμε καταρχήν να κάνουμε με την κατηγορία του αποθέματος. Ε, στα αριστερά λοιπόν βλέπουμε τα αποθέματα σε, στη, σε κατάσταση 2 ή 3 σε ό,τι αφορά ε, την αποκατάστασή του, Έχουμε γύρω στα 100 δηλαδή ήδη που περιλαμβάνονται ε, σε αυτή την κατηγορία και εδώ λοιπόν δίνουμε ε, συμβουλές με βάση τα στις στρατηγικές ή τα σχέδια διαχείρισης της αλίας εφόσον υπάρχουν και εφόσον τα εν λόγω σχέδια αξιολογηθούν ως συμβατά με την προληπτική ε, προσέγγιση και έχουν συμφωνηθεί από όλους τους ε, ε, συναποφασίζονται σε ό,τι αφορά το σχέδιο διαχείριση, τόσο εγκρίνονται. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποια αντίρρηση από τους συναποφασίζοντες ή δεν υπάρχει σημαντότητα με την προαιρετική προσέγγιση, τότε βασιζόμαστε στην προσέγγιση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης του MSY. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατηγορία 3 που έχουμε γύρω στα 80 θέματα όπου έχουμε δηλαδή παρατηρούμε ερευνητικά κάποιες ε, δειγματοληπτικές δηλαδή, έχουμε δειγματοληπτικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των αποθεμάτων, δίνουμε συμβουλές με βάση την προληπτική προσέγγιση και όχι τις μέγιστες βιώσιμες απόδοσεις, όπου δηλαδή λαμβάνονται ακριβώς υπόψη, ή, λαμβάνεται υπόψη η δυναμική εξέλιξη του αποθέματος και δίνονται συμβουλές με βάση αυτή την εξέλιξη. Είτε δηλαδή είναι αύξουσα ή φθήνουσα η ε, εξέλιξη του αποθέματος και πάντοτε Δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη μας και φροντίζουμε ή ε, αξιοποίηση των αποθεμάτων, η αλία να γίνεται με βάση την προληπτική προσέγγιση. Υπάρχουν τώρα μία σειρά από διαφορετικά σενάρια, όπω είπαμε, τα οποία υπολογίζουμε και τα οποία βασίζονται στου διάφορου κανονισμού οι οποίοι ε, βρίσκονται Ε, για παράδειγμα, εδώ στα αριστερά βλέπετε ε, την, ε, το πολιετές σχέδιο διαχείρισης ε, για τα βενθοπελαγικά είδη της Βορειοθάλασσας. Έχουμε λοιπόν εκεί τους διάφορους στόχους που οι προβλέπονται μέσα στο σχέδιο πολιτείου διαχείρισης. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την Ισλανδία, εκεί η Ισλανδία θα προβλέπει σχέδια διαχείρισης των διαφορετικών αποθεμάτων και ακριβώ οι συμβουλέ που εμεί θα παράσχουμε ω ISIS θα βασίζονται στο σχέδιο διαχείριση τη Αλία που θα έχει εκπονήσει η Ισλανδία. Όπως σας ε, είπα τώρα, όλες οι στρατηγικές ε, διαχείρισης της αλίας, επί των οποίων νομοδοτή δίνει συμβουλές ε, το ISIS, εξετάζονται με βάση προσωμιώσεις. Και πάντοτε εξετάζουμε μόνο τις, τις προοπτικές με βάση την προληπτική προσέγγιση. Δηλαδή εξηγούμε στις διάφορες οργανώσεις ότι υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικές δυνατότητες και σενάρια τα οποία εξετάζουμε και υπάρχουν κάποιοι ε, διαφορετική αν θέλετε αντικρουόμενη στόχη. Δηλαδή τι θέλετε να έχετε καλύτερη βιομάζα, ε, θέλετε να έχετε υψηλότερα TAC ή δηλαδή στα επιτρεπόμενα αλλιεύματα ή θέλετε να διατηρήσετε πολύ χαμηλό τον κίνδυνο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο απόθεμα. Ε, εδώ για παράδειγμα βλέπετε στα αριστερά ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη δηματοληψία σε σχέση με τον γάδο της Βορείου Θάλασσας. Βλέπουμε λοιπόν την ιστορική εξέλιξη του συγκεκριμένου αποθέματος και μετά εκεί που βλέπετε την κάθετη γραμμή ε, σταματάει η λήψη των στοιχείων και από εκεί και μετά λοιπόν το υπόλοιπο είναι η ε, πρόβλεψη που κάνουμε με βάση ακριβώς ε, τα στοιχεία που έχουμε και την ιστορική εξέλιξη. Κάνουμε λοιπόν μια προσωμείωση σε ό,τι αφορά τη μελλοντική εξέλιξη του συγκεκριμένου αποθέματος με βάση τις έρευνες που κάνουμε και ούτω καθεξής. Και από εκεί και μετά λοιπόν εξετάζουμε το πώς ακριβώς η εξέλιξη του εν λόγω αποθέματος εξελίσσεται μέσα στον χρόνο με βάση συγκεκριμένου στόχου και συγκεκριμένα σημεία ενεργοποίηση τα οποία έχετε προβλέψει στο, στο σχέδιο διαχείρισή σα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη θνησιμότητα στο 0,2-0,3 ή για παράδειγμα την θνησιμότητα που μπορεί να βρίσκεται στου 500-800.000 ετών ή οτιδήποτε άλλο. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία κάνουμε τι διάφορε προσωμιώσει έτσι ώστε οι αρμόδιοι για τα εν λόγω σχέδια διαχείριση να αποφασίζουν τι είδου είδου αλληλεία και σε ποιο βαθμό την επιθυμούν στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων ε, σχεδίων διαχείρισή του. Ε, τώρα, ποιο είναι ο κανόνα σε ό,τι αφορά τι συμβουλέ του ISIS, που αποτελεί ουσιαστικά τη βάση για τι τις περισσότερε από τι συμβουλέ που δίνουμε, είναι το εξή. Θα πρέπει να μεγιστοποιείται η μακροπρόθεσμη μέση απόδοση ταυτόχρονα όμως προστατεύοντα ε, το χαμηλότερο επίπεδο της από αποθέματος αναπαραγωγή. Ε, δηλαδή δεν θέλουμε να φτάσει το απόθεμα σε τόσο χαμηλά επίπεδα έτσι ώστε να μην είναι πλέον σε θέση να αναπαραχθεί. Άρα λοιπόν αυτό ο κανόνα σε ό,τι αφορά στι συμβουλέ μα έχουμε θέσει ένα συγκεκριμένο σημείο ενεργοποίηση το οποίο λέγεται B-Trigger και είναι ακριβώ σε ό,τι αφορά τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Εφόσον λοιπόν ένα απόθεμα βρίσκεται πάνω από αυτό το MSY τότε μπορεί να λαμβάνει χώρα η αλίευση στο επίπεδο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Και σε περίπτωση δηλαδή πολυετών ε, σχεδίων ε, αλληλείας, ε, για παράδειγμα στη Βόρειο Θάλασσα, στη Βαλτική ή αλλού, έχουμε και κάποια φάσματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν δύο διαφορετικά MSY. Το ανώτατο για παράδειγμα, ε, μέχρι απόδοσης και το χαμηλότερο. Και από εκεί και μετά, εάν φτάσει να πέσει κάτω από το ε, από αυτό το σημείο αναφορά σε MSY, δηλαδή το σημείο ενεργοποίηση και αρχίζει να κατευθύνεται προ το Bill lim δηλαδή το σημείο που είναι επικίνδυνο πλέον για την αναπαραγωγή, έχουμε την γραμμική ε, μείωση της ε, ε, θνησιμότητας ακριβώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία, δηλαδή το B3 και το B-lim. Αν βρισκόμαστε κάτω από την B-lim, εξετάζουμε την κατάσταση του αποθέματο και βλέπουμε μπορούμε να βράχει πρόθεσμα να αποκαταστήσουμε το απόθεμα ώστε να βρεθεί πάνω από το B-lim, για παράδειγμα στο 2021. Θέτοντας δηλαδή ένα συγκεκριμένο στόχο σε ό,τι αφορά την εθνισμότητα από την αλληλεία. Εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε, αν δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε αποκατάσταση ε, βράχη πρόθεσμα πάνω από το πιλίμ, τότε η συμβολή από την πλευρά του ΆΣΙΣ θα είναι μηδενική αλία, απαγόρευση της αλίας για το συγκεκριμένο απόθεμα. Και έχουμε δώσει τέτοιου είδου συμβουλέ ε, για μια σειρά από είδη από θέματα δηλαδή ε, σε σχέση με τα οποία δεν ήταν ακριβώς δυνατό να υπάρξει βράχη πρόθεσμη αποκατάσταση του αποθέματος έτσι ώστε να βρεθεί πάνω από τον πυλήμ. Εκεί δηλαδή χρειάζεται να προβλεφθούν συγκεκριμένα σχέδια σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του αποθέματος και σε σχέση με αυτά τα σχέδια ε, το ISIS δίνει και πάλι συμβουλές. Δεν υπάρχουν κάποιο, ε, κάποια τέτοια σχέδια αυτή τη στιγμή, αλλά τι θα περιλάμβανε ένα τέτοιο σχέδιο αποκατάστασης δηλαδή του αποθέματος. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ε, συγκεκριμένη ε, προοπτική για 10 χρόνια ή οτιδήποτε άλλο, για μια μισή γενιά των χθείων, οτιδήποτε άλλο, όπου θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνε ως προς το πώ ακριβώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος τη αποκατάσταση. Τώρα, όλα τα σημεία αναφοράς έχουν και ένα ανώτατο όριο, έτσι ώστε δηλαδή πάντοτε να βρίσκονται εντό της προαιρετικής προσέγγιση. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε ακριβώς την ε, αλληλεία στα επίπεδα τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση να μην αρχίσει να μειώνεται και προ το billing το συγκεκριμένο απόθεμα. Θα σα δώσω τώρα ένα παράδειγμα ω προ το. Ε, για το και έχουμε για παράδειγμα εδώ ένα παράδειγμα και είναι ενδιαφέρον γιατί ε, στα, γύρω στις 50, 40 με 50 χιλιάδες ετώνους είχαμε στη δεκαετία του 70 και του 80 με αποτέλεσμα να αρχίσει να μειώνεται σταθερά το συγκεκριμένο απόθετα, απόθεμα και αν, δείτε το ε, MSC ε, είδαμε από τους 100.000 ετώνους να μειώνεται Ε, και ε, συνεχίστηκε αυτή η μείωση, είναι, πρόκειται για το Μερλούκιο εδώ, ε, και μετά τέθηκε σε ισχύ ένα σχέδιο αποκατάστασης το οποίο πράγματι οδήγησε σε σημαντική μείωση της νησιμότητας από την αλληλεία του εν λόγω αποθέματος και είδαμε να, είναι πράγματι, να γίνεται βιώσιμη πλέον αυτή να γίνεται βιώσιμη ή εν λόγω αλληλεία μέσω αυτής της μειωμένης μέσα στην επόμενη λοιπόν δεκαετία άρχισε να μειώνεται πολύ σημαντικά η θνησιμότητα και βρίσκεται πάνω πλέον το επίπεδο από το ε, μέγιστο βιώσιμης απόδοσης και κατά συνέπεια η βιομάσα του αποθέματος αναπαραγωγής έχει ανταποκριθεί και βρισκόμαστε πλέον στα 330.000 ε, τόνους ως ε, βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής για τον Μερλούκιο. Και βλέπετε λοιπόν ε, ότι τα επίπεδα σε ό,τι αφορά την προσθήκη των νέων εχθρών, δηλαδή την αναπαραγωγή, δεν ε, έχουν μεταβληθεί ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν η ανταπόκριση του αποθέματο οφείλεται ακριβώ στη μείωση τη νησιμότητα. Ακριβώ δηλαδή με τη μείωση τη αλληλεία καταφέραμε την αποκατάσταση του αποθέματο. Βλέπετε εδώ λοιπόν τα αλλιεύματα ε, το 2018, 96.000 τόνοι και η συμβουλή δηλαδή που δώσαμε είναι ε, ε, λίγο υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2018 ε, και όταν κάνουμε κάποιες προβλέψεις εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αναλύσεις ό,τι αφορά την εθνισμότητα. Για το παράδειγμα το 2019 κάνουμε και μία πρόβλεψη και με βάση αυτή την εθνισμότητα κάνουμε μία πρόβλεψη ή μάλλον κάνουμε την πρόβλεψη του αλλιεύματος για το 2020 με βάση την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, δηλαδή εκείνο το επίπεδο αλλιεύματος και δίνουμε ακριβώς και κάνουμε αυτή την πρόβλεψη για 104.000 τόνους. Πράγμα το οποίο οδηγεί σε μια βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής ε, της τάξης των 263.000 τόνων για το 2021 που, μιλά, που οδηγεί σε μείωση κατά 50% αυτού του αποθέματος του, της βιομάζας δηλαδή αναπαραγωγής. Μετά, για τα ε, δυτικά έδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάποια ε, φάσματα για το FMSY, για το χαμηλότερο δηλαδή. Θα είναι 76.000 τόνοι, ενώ το ανώτερο είναι 147, ε, με 148.000 τόνους. Αυτή είναι λοιπόν η επιστημονική συμβουλή. Θα σας διακόψω, λέει ο Πρόεδρος και όποιος θέλει να παρέμβει παρακαλώ να πάρει το λόγο. Για να σας πω το εξής. Όταν ε, τίθεται το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ασκούν ε, κριτική στην Επιτροπή και λένε ότι βασίζεστε σε επιστημονικές συμβουλές, αλλά ως Επιτροπή παίρνετε μόνο το, ε, το, χαμηλότερο, το μέγιστο δυνατό όριο, ενώ οι επιστήμονες δίνουν ένα εύρος από ελάχιστο σε κατώτατο όριο. Σα ρωτώ λοιπόν την άποψή σας. Ένας πολιτικός, όταν ένα επιστήμονα του δίνει μία πρόταση με, με ένα εύρο από χαμηλότερο σε ανώτερο όριο, ποιο θα πρέπει να επιλέξει. Παίρνει το λόγο η συνάδελφος για να πει ότι έχουμε ένα benchmark για τη σύγκριση. Για τη σύγκριση. Συμφωνείτε με αυτό? Όχι ακριβώς, ε, λέει ο κύριος Κον θα σας εξηγήσω. Ο λόγος για τον οποίο δίνουμε ένα εύρος, δύο τιμές, μία ανώτερη και μία κατώτερη, είναι γιατί προβλέπεται στην νομική τεκμηρίωση, στο πολιετές σχέδιο, το οποίο αποτελεί μέρος της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Το δίνουμε γιατί μας το ρωτάτε. Εσείς μας ζητάτε να δώσουμε εύρος και γι' αυτό δίνουμε εύρος. Το πάνω μέρος του φάσματος αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο οι ορισμένε προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πολιετές σχέδιο, οι οποίες μάλιστα είναι και πολύ αυστηρές. Και μπορώ να σας τις αναφέρω αν θέλετε. Το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα δεν έχει τεθεί με βάση το ανώτατο όριο εξ όσο γνωρίζω. Δηλαδή παρόλο που υπάρχει ένα φάσμα, ένα εύρος για τη Βαλτική θάλασσα και τη Βόρεια θάλασσα, ήδη δύο χρόνια για τη Βαλτική, το άνω κομμάτι του φάσματος αυτού δεν έχει χρησιμοποιηθεί γιατί η επιστημονική επιχειρηματολογία ε, θεωρεί ότι δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθεί το πάνω μέρος του φάσματος. Το ανώτερο όριο του φάσματος είναι η τιμή του FMS για τις περισσότερες συμβουλές που δίδουμε, δηλαδή αυτό υιοθετούμε. Μερικές φορές ε, δεν ταιριάζουν σωστά ε, τα νούμερα στις συμβουλές του ISIS. Για παράδειγμα, για τον ε, Πακαλιάρο Μερλούκιο της Βόρειας Θάλασσας, Έχουμε αποθέματα από το κόλπο τον Βυσκαϊκό μέχρι την Βόρεια Θάλασσα και το Σκάγκερακ. Έχουμε διάφορες τιμές και έχουμε τέσσερα διαφορετικά μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Μερικέ φορέ καλή σύγχυση, επικρατεί σύγχυση γιατί έχουμε ένα μέγιστο επιτρεπόμενο αλλιεύμα για μία περιοχή από αυτή την τεράστια περιοχή από τον κόλπο το Βυσκαϊκό μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα και τη θάλασσα του Σκάγκερακ για το ίδιο ψάρι. Και υπάρχει λάθος αντιστοιχεία δηλαδή και παρανόηση. Ε, η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι για την πλειονότητα των ηχθειαποθεμάτων τηρεί τις επιστημονικές συμβουλές. Ο Πρόεδρος. Άρα αυτή είναι η αξιολόγησή σας. Το πιστεύετε. Απάντηση. Νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί πολύ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ξεκινούσαμε δίναμε απλά έτσι συμβουλές και υπήρχε μια συζήτηση. Αλλά τώρα με την μεταρρύθμιση της κοινή ελιευτικής πολιτικής και την μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση είναι πολύ πιο αυστηρές, αυστηρό το πλαίσιο και ε, υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια να ε, τηρηθούν ε, τα, ε, τα επιστημονικά ε, πορίσματα. Μιλούμε για 104.000 τόνους εδώ σε σχέση με το ερώτημά σας. Αυτό είναι το εύρος. Το, έχουμε ήδη λάβει υπόψη αυτό που λέτε. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ευχαριστώ, συνεχίζω. Επομένως, διαχείριση με βάση το οικοσύστημα. Όπως είπα και εξ αρχής, δίνουμε συμβουλές για 240 ηχθη από θέματα, ξεχωριστά για το καθένα. Αλλά πρέπει να δώσουμε και συμβουλές για το ευρύτερο οικοσύστημα. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε συμβουλές για το πώς θα διαχειριζόμαστε την ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει αντίκτυπο στο εκάστοτε οικοσύστημα. Και για να το πράξουμε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αλληλευτική πίεση στο κάθε ήχθη απόθεμα, αλλά και συλλογική πίεση σε όλα τα ήχθη αποθέματα και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα πρέπει να προσέχουμε το καλό, την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, η καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, GES το αρτικόλεξο, χρησιμοποιείται στην οδηγία και διάφοροι στόχοι έχουν ε, καθοριστεί με βάση αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη την καλή κατάσταση, για την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος όχι μόνο τα αχθιοποθέματα αλλά και άλλα στοιχεία του ευρύτερου θαλασσίου περιβάλλοντο. Θέλουμε να, έχουμε, να πετύχουμε αυτή την καλή περιβαλλοντική κατάσταση, την αηφόρο χρήση, να βελτιστοποιήσουμε τα ωφέλη ε, που ε, θα βοηθήσουν την κοινωνία να επιδιώξει τους στόχους της. Θέλουμε να έχουμε την περιφερειοποίηση, την περιφερειακή διάσταση και σωστά αντισταθμίσματα. Ε, το αν θα είναι τα αλλιευτικά σκάφη μικρά ή μεγάλα δεν είναι θέματα που απασχολούν την επιστήμη. Η επιστήμη μπορεί να συμβουλεύσει και να βοηθήσει, αλλά τελικά η κοινωνία είναι αυτή που θα πάρει τις αποφάσεις. Το βασικό όμως είναι να ε, πλαισιώσουμε και να βοηθήσουμε το οικοσύστημα έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Έχουμε πολύ διαφορετικές ε, περιφέρειες και περιοχές γύρω από την Ευρώπη στο Βορειοατλαντικό ωκεανό Κάνουμε μία επισκόπηση αναλυτική για κάθε μία από αυτές τις περιφέρειες ή περιοχές και κάποια από τα αποτελέσματα θα σας τα παρουσιάσω εντός ολίγου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των πόρων και την βιοπικιλότητα, τους στόχους δηλαδή για τη διατήρηση αυτών. Εμείς ε, συμβουλεύουμε και την ΙΑΦΚ, την ε, ε, Λευτική Επιτροπή για το Βορειοατλαντικό Ωκεανό και απαντούμε σε διάφορα αιτήματα από την ΕΑΦΚ και από την ΟΣΠΑΡ, την Επιτροπή Όσλο Παρισιού. Και ε, οι δύο επιτροπές, η ΝΕΦ και η ΟΣΠΑΡ, συνεργάζονται και προσπαθούν να μεριμνήσουν για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε περιοχές που ε, εκτείνονται πέραν της ε, ευρωπαϊκής ή εθνικής δικαιοδοσίας. Παρέχουμε συμβουλές και στη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και στη Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΙ για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η DG ΜΑΡΕ ασχολείται με την κοινή αλληλευτική πολιτική και η DG ΕΝΒΙ ασχολείται με τις οδηγίες για τους βιοτόπους ε, και για τα πτηνά και για το στρατηγικό πλαίσιο για το θαλάσσιο περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση οι συμβουλές που παρέχουμε πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια, συνοχή, να συνάδουν με τους στόχους και να γεφυρώνουν τα παραδείγματα πάνω στα οποία στηρίζονται. Ε, κάθε φορά υπάρχουν κάποια περίπλοκα ζητήματα, κάποια αντισταθμίσματα ε, και όταν παρέχουμε συμβουλές πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη για να φτάνουμε σε ένα σωστό σημείο ισορροπίας. Θέλουμε οι συμβουλές μας να μπορούν να είναι λειτουργικές. Άρα μας ενδιαφέρει το πώς ένα δυναμικό οικοσύστημα επηρεάζει την αλία, τα αλλιευτικά αποθέματα. Όλοι γνωρίζουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και αυτό έχει τον αντίκτυπό του στα αποθέματα και στη δυναμική αυτών των τελευταίων. Εξετάζουμε τον αντίκτυπο της αλλιευτικής δραστηριότητας στο οικοσύστημα και παρέχουμε στοιχεία. Άρα εξετάζουμε το πόσο αντίκτυπο έχει η αλευτική δραστηριότητα με τράτες οι οποίες φτάνουν μέχρι το πυθμένα ε, της θάλασσας, στο εκάστοτε οικοσύστημα και στα ηχθή αποθέματα. Επίσης υπάρχει ανταγωνισμός για το διάστημα από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες και αυτό έχει αντίκτυπο στον ωκεανό. Βλέπουμε λοιπόν ε, τις συνέπειες που έχουν οι, κάθε, οι στόχοι διαχείρισης. Όπου χρειάζεται λαμβάνουμε υπόψη αλλαγές στην παραγωγικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηχθιαποθέματα. Μιλούμε για ε, την ανάπτυξη, τη φυσική θνησιμότητα, όλα μεταξύ άλλων, όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη στην αξιολόγηση που κάνουμε για τα ηχθή αποθέματα, για τις προβλέψεις μας και για τα σημεία αναφοράς που θα εδραιώσουμε. Βλέπουμε τις αλλαγές και τις επικαλύψεις που μπορεί να υπάρχουν στην κατανομή των ηχθή αποθεμάτων και εξετάζουμε εναλλακτικές ε, ε, στρατηγικές διαχείρισης, ε, διαφορετικά σενάρια παραγωγικότητας. Αυτό το κάνουμε όταν αξιολογούμε τις διαχειριστικές στρατηγικές, όταν μας ρωτούν πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα ένα ηχθειοπόθεμα, βλέπουμε τα διαφορετικά καθεστώτα και εξετάζουμε πώς θα ανταποκριθεί το διαχειριστικό σχέδιο σε περίπτωση που θα επέλθει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο συγκεκριμένο απόθεμα. Κατά πόσο δηλαδή η στρατηγική διαχείριση έχει και αναλλακτικά σενάρια και προβλέπει για διάφορες ε, εξελίξεις διαφορετικές. Τώρα, σε σχέση με τα παραλιεύματα ή τα παράπλευρα λιεύματα, ε, τα μετράμε, κάνουμε αναφορά στη συχνότητά της, στη συχνότητα εμφάνισής τους και τον αντίκτυπο αυτών και βλέπουμε τον αντίκτυπο της αλλιευτικής δραστηριότητας και των λοιπόν υπηρεσιών στα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, τα VME. Συνθέτουμε πληροφορίες, πληροφορίες και κάνουμε τη σύνοψη όλων αυτών για να έχουμε μια συνοπτική απεικόνηση και ολοκληρωμένη ε, για την κατάσταση του συγκεκριμένου ηχθιαποθέματος στην εκάστοτε οικολογική περιοχή. Προσπαθούμε η, η αλληλεία να μπαίνει σε ένα πλαίσιο ευρύτερο όπου θα την εξετάζεται συνολικά μαζί με τις λοιπές θαλάσσιες δραστηριότητες και πιέσεις που ασκούνται στις θάλασσες ή στους ωκεανούς γιατί θέλουμε τελικά να καθορίσουμε ε, τις πιέσεις σε μια περιοχή, σε ένα οικοσύστημα από το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θέλουμε ε, να έχουμε πληροφορίες και μεθόδους έτσι ώστε να καθορίσουμε ότι μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή είναι οικολογικός ή βιολογικός σημαντική και άρα μπορεί να απειλείται ή να μην απειλείται. Θέλουμε να παρακολουθούμε τις τάσεις στα διάφορα είδη, τη βιοπικιλότητα και τη δομή του οικοσυστήματος. Έτσι πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στο να γίνει καλύτερη αξιολόγηση των επαπειλούμενων ε, ειδών ή των ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση ή βιοτόπων που κινδυνεύουν επίσης με εξαφάνιση και παρακολουθούμε και τη συχνότητα εμφάνισης των χωροκατακτητικών ειδών. Ε, έχουμε ομάδες αξιολόγησης των οικοσυστημάτων που εξετάζουν ε, ε, από κοινού όλους τους στόχους διαχείρισης. Προσπαθούμε να έχουμε εργαλεία για να συγκρίνουμε τις διάφορες δράσεις και τα διάφορα αντισταθμίσματα και θέλουμε τη δέσμευση των ε, εμπλεκόμενων φορέων ότι θα δεσμευτούν δηλαδή ότι θα αξιοποιήσουν τις μεθόδους, τις ιδέες που τους παρέχουμε και θα έχουν υπόψη του τις συνέπειες. Θέλουμε δηλαδή οι συμβουλές μας να έχουν πρακτική εφαρμογή και να δούμε τον αντίκτυπο των θετικό των συμβουλών μας ε, στην κατάσταση του πυθμένα, στο στρατηγικό πλαίσιο και στην μεικτή αλλιευτική δραστηριότητα. Δημοσιεύουμε λοιπόν όλες αυτές τις συμβουλές όπως σας είπα, για πάνω από 240 ήχθη αποθέματα. Εξετάζουμε την επιρροή θεωρούμε ότι οι συμβουλές μας επηρεάζουν τη δυναμικότητα ενός οικοσυστήματος. Έχουμε σταματήσει να εξετάζουμε, το, να δίνουμε έμφαση στο κάθε ηχθιαπόθεμα ατομικά. Θέλουμε να έχουμε μια πολύ πιο συνολική προσέγγιση, να εξετάζουμε το οικοσύστημα στο σύνολό του και μάλιστα να εξετάζουμε και το σύνολο της αλληλευτικής δραστηριότητας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου θα λάβουμε υπόψη και την υπόλοιπη ανθρώπινη δραστηριότητα, ανθρωπογενή δραστηριότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη λυπή πίεση που ασκεί ο άνθρωπος στο εκάστοτε ε, περιβάλλον. Και ε, καταλήγουμε στον αντίκτυπο της αλληλευτικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο οικοσύστημα. Όλες λοιπόν αυτές οι συμβουλές παρέχονται και μπορεί κανείς να τις κατεβάσει από την ε, ιστοσελίδα μας. Εδώ ε, βλέπετε κάποιες από τις περιοχές στην Αλία, στην Κελτική θάλασσα, έχουμε κάποιες αναλογίες, κάποια ποσοστά. Έχουμε εκεί τις περιοχές όπου οι τράτες έχουν αντίκτυπο στον πυθμένα και στο βυθό. Βλέπετε ε, τα hot spot, εκεί όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος αντίκτυπος. Με τα κινητά εργαλεία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θα πει κινητά εργαλεία. Αλληλεία για αρχαρίους. Λοιπόν, κινητά εργαλεία είναι οι τράτες διαφόρων ειδών, δοκότρατες, πελαγικές και τα στατικά εργαλεία είναι τα δίχτυα που ρίχνουν. Δηλαδή, κινητά εργαλεία είναι οι τράτες οι διάφορες, τις οποίες σέρνει πίσω του το σκάφος καθώς προχωράει. Ενώ στατικά εργαλεία είναι τα δίχτυα που ρίχνει και η τράτα που ρίχνει και μαζεύει σε συγκεκριμένο σημείο. Βλέπετε ότι στη θάλασσα της Κελτικής έχουμε φόρτωση περίπου ενός εκατομμυρίου τόνου ηχθιαποθεμάτων από τα μέση της δεκαετίας του 80. Ο πρόεδρος, ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διαφάνεια. Βλέπετε, δείχνετε εδώ ότι υπάρχει αντίκτυπο στο πυθμένα, αλλά αυτό μας ανησυχεί. Βλέπω ένα hot spot, ένα κόκκινο σημείο, δηλαδή στα ανατολικά της Ιρλανδίας. Μιλούμε για την καραβίδα. Και εγώ ήμουν σε αυτό το λιμάνι, το Κικίλ, πριν από λίγες εβδομάδες και είδα ότι βγάζουν πολλά χρήματα από τις καραβίδες, τις οποίες, τις πολλούν στην υπηρετική αγορά. Είναι ένα λιμάνι δηλαδή που ευημερεί. Όμως εσείς το χάρτη το έχετε κόκκινο. Αυτό είναι κακά νέα για το μέλλον της καραβίδας ή είναι βιώσιμο και για την καραβίδα και για την οικονομική δραστηριότητα στο λιμάνι. Για αυτή την περίπτωση γίνεται αξιολόγηση του αποθέματος. Ε, σύμφωνα με την αξιολόγηση, πέρσι η καραβίδα αλλιευόταν με βιώσιμο τρόπο. Όμως, τι αντίκτυπο, ε, ποιος είναι ο αντίκτυπος με τα άλλα είδη που αλλιεύονται παράλληλα με την καραβίδα. Μιλούμε για τα παράπλευρα αλλιεύματα, τα οποία δεν αλλιεύονται βιώσιμα. Όπως το προσφυγάκι και εξετάζουμε και τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα κινητά εργαλεία στον, πυθε... πυθμένα. Πώς το διαχειριζόμαστε αυτό, αναστέλουμε την ε, αλίευση της καραβίδας ή πρέπει να βρούμε άλλες περιοχές όπου ε, θα διαβεί το προσφυγάκι και θα τις ανακηρύξουμε περιοχές ευπαθείς για να τις προστατεύσουμε εκεί και να επιβιώσει αυτό το είδος εκεί. Όλα αυτά εξαρτώνται λοιπόν από την εξέτασή μας και την αξιολόγησή μας. Προσπαθούμε δηλαδή να ταιριάξουμε αυτές τις καταρκεσματισμένες πληροφορίες για να έχουμε ένα τελικό σενάριο του κατά πόσο η ελευτική δραστηριότητα είναι βιώσιμη ή όχι. Εδώ βλέπετε μία επισκόπηση πάλι στην Κελτική θάλασσα για την θνησιμότητα αλλά και για την βιομάζα ε, της οτοκίας για όλα τα βυνθοπελαγικά είδη. Η μαύρη γραμμή είναι η θνησιμότητα. Κατά μέσο όρο βλέπετε ότι η τάση είναι πτωτική προς την οριζόντια γραμμή που είναι η γραμμή που προκύπτει από το στρατηγικό πλαίσιο και την βιώσιμη διαχείριση. Άρα η τάση είναι θετική συνολικά, αλλά κάποια ηχθιαποθέματα ξεχωριστά ατομικά παρουσιάζουν πολύ, μεγάλη, ε, πολύ ψηλή θνησιμότητα. Αυτά τα συγκεκριμένα. Ενώ συνολικά κινούμαστε προς μια θετική κατάσταση. Ορισμένα ηχθιαποθέματα μάλλον γίνεται αντικείμενο ακόμα ε, εντατικής υπεραλίευσης και υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε τη βιομάζα, την οτοκία και σε σχέση με τη μέγιστη ε, απόδοση, τη βιώσιμη. Βλέπετε ότι κατά μέσο όρο υπάρχει άνοδος, όμως ε, κάποια αποθέματα παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν ε, ξαναγεννιούνται αρκετά. Δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο δηλαδή οτοκίας. Η πάνω διαφάνεια έχει να κάνει με τη θνησιμότητα και η κάτω διαφάνεια με την γεννητικότητα, με και βλέπουμε λοιπόν ότι οι τάσεις είναι θετικές, αλλά κατά μέρος με μονομένες περιπτώσεις είναι προβληματικές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τους διαφόρους στόχους που δείχνουν το επίπεδο της θνησιμότητας. 59 ηχθιαποθέματα που ε, δεν είναι γνωστό το καθεστώς σε σχέση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, όμως στο κάτω μέρος της διαφάνειας βλέπετε τα το ετήσια αλλιευτική δραστηριότητα και αντιστοιχεί σε πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής αλλιευτικής δραστηριότητας. 16 ηχθιαποθέματα είναι στο κόκκινο, δηλαδή γίνονται αντικείμενο εντατικής υπεραλίευσης και Αυτά προέρχονται από την υψηλότερη πλειοψηφία των εκφορτώσεων στην οικοπεριοχή. Κάποια άλλα ε, γίνονται αντικείμενο βιώσιμης εκμετάλλευσης και αυτά τα αποτελέσματα έχουμε όταν κοιτούμε τη θνησιμότητα. Όταν δούμε λοιπόν όμως την βιομάζα και την οτοκία, εκεί η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Ε, το μεγαλύτερο μέρος είναι πράσινο σε σχέση με τις εκφορτώσεις. Δηλαδή, άρα βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της αλίευσης γίνεται από βιώσιμα ως σπόρους με υψηλό ε, και βιώσιμο ποσοστό και επίπεδο βιομάζας. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη συγκριτική μελέτη για να ε, καταλήξουμε σε συγκεκριμένες πληροφορίες και να έχουμε τη γενικότερη εντύπωση του πώς θα πηγαίνει η συγκεκριμένη οικολογική περιοχή. Και στην επισκόπηση για το οικοσύστημα, π.χ. στη Βόρεια Θάλασσα, Έχουμε συγχωνεύσει τις ομάδες εργασίας. Η κάθε ομάδα εργασίας ασχολείται με τη χαρτογράφηση της εκάστοτε ανθρώπινης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Εντοπίζει ποιες πιέσεις ασκούνται στην εκάστοτε περιοχή, πόσες είναι αυτές και ποιο αντίκτυπο έχουν σε κάθε μία από τις συνιστώσεις, σε κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Και βλέπουμε έτσι τις προτεραιότητες. Ποιε θα πρέπει να είναι οι περιοτεραιότητες. Θα πρέπει η διαχείριση της οικολογικής ε, περιοχής να ασχοληθεί περισσότερο και κατά προτεραιότητα με την αλληλευτική δραστηριότητα ή με την ε, δραστηριότητα των βυθοκορήσεων και της εξόρυξης ε, και των αντλήσεων των πετρελαϊκών ή άλλων πόρων. Εδώ βλέπουμε τις εγκαταστάσεις για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα και έχουμε και τη βασική παραγωγικότητα του οικοσυστήματος. Ο χάρτης αυτός μας δείχνει την πρωτογενή παραγωγικότητα στην Βόρεια Θάλασσα. Με κόκκινο είναι τα σημεία όπου έχουμε υψηλή ε, πρωτογενή παραγωγή τα τελευταία χρόνια. Και βλέπετε ότι σε βάθος χρόνου μειώνεται αυτή η πρωτογενής παραγωγικότητα στη Βόρεια Θάλασσα, διότι τα διάφορα νητρικά και ε, φωσφορούχα ε, ουσίες μπαίνουν ε, μπαίνουν στον ωκεανό από, την, από τα ποτάμια τα διάφορα που εκβάλλουν και έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα των υδάτων του ωκεανού. Άρα μειώνονται τα νητρικά. Ναι, αυτό είναι καλό. Δεν είναι και τα φωσφορικά άλατα. Καλό είναι γιατί δεν μολύνουμε τους ωκεανούς. αλλά έχουμε μείωση πρωτογενής, πρωτογενής παραγωγικής δραστηριότητας και αλλαγή της σύστασης. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει από τους ε, ε, πόρους ε, της γης, αναλόγως με τα είδη κάποιο είδος θα ωφεληθεί δηλαδή και κάποιο άλλο είδος θα ε, έχει πρόβλημα. Δεν τα κάνετε εύκολα για τους πολιτικούς. Είναι όντως περίπλοκο το θαλάσσιο περιβάλλον. Δεν είναι μία και απλή λύση. Να σας κάνω μία σύνοψη τώρα όλων όσων είπα. Είμαστε μία παγκόσμια οργάνωση για τη θάλασσα. Ε, δίνουμε αμερόληπτα στοιχεία ε, στους πολιτικούς, ε, που βασίζονται σε επιστημονικά, συμβουλές που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Οι συμβουλές του ΆΙΣΙ συνάδει με διάφορους στόχους πολιτικής ε, που θέτονται θετικώς όπως η αρχή της προφύλαξης, η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, η διαχείριση με βάση το οικοσύστημα και τα χαρακτηριστικά του και όλα αυτά αναφέρονται ε, και στην κοινή αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνή νομοθεσία που υπάρχει και άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι μέλη του ISIS έχουν αντίστοιχες, αντίστοιχους ε, παράγονται οι συμβουλές. Είναι οι ενεργοί εμπειρογνώμονες, 1500 ενεργοί εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται 1500 ενεργοι εμπειρογνώμονε που δραστηριοποιουνται εντο του ISIS. Εμείς δεν τους πληρώνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, Πολύ λίγοι από αυτούς που συμμετέχουν στις δραστηριότητε μας πληρώνονται. Βασικά πληρώνονται από τα δικά τους Ινστιτούτα για να συνεισφέρουν στο έργο του ISIS. Δεν έχουμε απεριόριστους πόρους. Γιατί θεωρούν ότι είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο και αυτό ευθυγραμμίζεται με τους στόχους των ε, Ινστιτούτων τους ή των οργανώσεών τους και των χωρών μελών από ε, τις οποίες προέρχονται. Άρα η ατμομηχανή ουσιαστικά ε, του ISIS χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες μέλη του ISIS. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την επιστημονική κοινότητα που κάνει αυτό το ερευνητικό έργο μέσω ε, χρηματοδότησης. Η τελική συμβουλή ε, με συνένεση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ISIS Έχουμε εκεί 20 μέλη, ε, ένα χώρα, συν 5 ακόμα, 4 αντιπρόεδρους και ένα πρόεδρο. Η συλλογή των δεδομένων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να δώσουμε συμβουλές για την βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. Είναι κρίσιμο να έχουμε τις ροές αυτών των δεδομένων ε, που, και να τα λαμβάνει αυτά τα στοιχεία ο ISIS, τα χρησιμοποιεί πολύ σωστά, κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση όλων των δεδομένων που συλλέγονται. Είναι πάρα πολύ δαπανηρό να συλλέξουμε όλα αυτά τα δεδομένα, είναι πάρα πολύ δαπανηρό να κάνουμε μεγάλα, να χρηματοδοτούμε μεγάλα ερευνητικά σκάφη, ας πούμε, όπως αυτό που έχουμε το Celtic Explorer στην Κελτική. Και προσπαθούμε λοιπόν ε, όλα αυτά να συνεισφέρουν στην συμβουλή που δίνουμε βάση στοιχείων για μια βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. Γιατί χρησιμοποιούμε μοντέλα πληθυσμών στον ISIS για να δώσουμε μία εικόνα για την ιστορική εξέλιξη των νυχθιαποτευμάτων, να δούμε την θνησιμότητά του, την ε, βιομάζα της, ε, του αναπαραγωγικού αποθέματος ε, και την ανανέωση του πληθυσμού. Έχουμε ιστορικά στοιχεία για ό,τι συνέβη στο απόθεμα και κάνουμε μία πρόβλεψη για το μέλλον. Έχουμε σημεία αναφοράς που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουμε την κατάσταση του αποθέματος ε, αν είναι σε καλή κατάσταση, αν είναι σε κακή κατάσταση, ανάλογα με τα διάφορα σημεία αναφορά που έχουμε καθορίσει και κάνουμε μία βραχυπρόθεσμη ε, πρόβλεψη για να υπολογίσουμε διάφορα τάκ, μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα και οι βασικές συμβουλές που δίνουμε βασίζονται πάντα στους στόχους διαχείρισης εκείνων που μας ζητούν ε, συμβουλές για ε, τη διαχείριση των αποθεμάτων. Και κάνουμε και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για να αξιολογήσουμε τις ε, στρατηγικές διαχείρισης Βλέπουμε τι δούνε και λαβή να μας προσφέρει κάθε προσέγγιση για τη διαχείριση του αποθέματος και προσπαθούμε να πιέσουμε και να δημιουργήσουμε μία επισκόπηση για την αλληλεία και τα οικοσυστήματα και να συνοψίσουμε και να συγχωνεύσουμε και να αθροίσουμε τις γνώσεις που έχουμε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς δουλεύετε με τους αλείς για να συλλέξετε τα δεδομένα. Γιατί συχνά οι ψάδες μας λένε ότι οι εμπειρογνώμονες και οι επιστήμονες είναι στον κόσμο τους, δεν τους ακούνε κτλ. Το άκουσα πάρα πολλές φορές να το λένε αυτό. Κοιτάξτε, όταν είπατε ποιος είσαστε, είπατε ότι έχετε υπάρξει και αλίας. Ε, ψαρέψατε σε διάφορα κόντεξτ. Ας πούμε, κανένας δεν μπορεί να σας κατηγορήσει ότι είστε απλώς ένας καθηγητής που κάθεται στην καρέκλα του. Η σχέση με τους αλίες είναι περίπλοκη ανάμεσα στο, στους ε, τον κλάδο δηλαδή και τους επιστήμονες. Έχουμε προγράμματα ε, με δειγματοληψία των αποθεμάτων ε, σε όλες τις χώρες. εκατό της ε, αληφτικής δραστηριότητας παρατηρείται από επιστήμονες που παρατηρητούν και συλλέγουν δεδομένα και τα χρησιμοποιούμε για να τροφοδοτήσουμε τις αξιολογήσεις για το απόθεμα. Ένας τρόπος επαφής με, την, με τον κλάδο είναι αυτός. Επίσης, έχουμε ε, εργαστήρια. Πρόσφατα έγινε ένα εργαστήριο. WK Cindy λέγεται, το τελευταίο που έγινε, που είναι ένα εργαστήριο το οποίο κοιτάζει πώς η επιστήμη και ο αληθικός κλάδος μπορούν να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά στο μέλλον ε, για τη συλλογή των δεδομένων και να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν οι αλήσει οι ίδιοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιστημονική διαδικασία και να το θεωρούν να τις νόμιμες αυτές ε, και μη προκατηλημένες πληροφορίες. Τα τελευταία τρία χρόνια οι μεγάλες οργανώσεις παραγωγών άρχισαν να προσλαμβάνουν επιστήμονες παύλα ψαράδες, οι οποίοι ε, συνεργάζονται με τους ψαράδες για τη συλλογή δεδομένων. Και ετοιμάζουμε και έρευνες για να βελτιώσουμε τη συλλογή των δεδομένων και τη δημιουργία στοιχείων. Και όταν υπάρχουν κενά ανάμεσα στα στοιχεία και στα δεδομένα, προσπαθούμε να υπάρξει συνεισφορά από τους αλληλείς ε, και αυτά τα στοιχεία τροφοδοτούν τα επιστημονικά προγράμματα. Επομένως, έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση σε ε, εθνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο ISIS. Επομένως, ε, λίγοι επιστήμονες είναι πάνω στα σκάφη. Φυσικά συνεργάζονται με τους καπετάνιους, έτσι. Πώς είναι η σχέση τους. Δεν φαντάζομαι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν κάποιον να τους αστυνομεύει. Υπάρχει νομική υποχρέωση, λέει ο μιλητή, που προβλέπεται σε ένα από τους κανονισμούς, δεν θυμάμαι ποιον. Τα σκάφη να δέχονται επιστημονικούς παρατηρητές. Είναι στον κανονισμό συλλογή δεδομένων ίσω. Υπάρχει νομική υποχρέωση που βαραίνει τα σκάφη. Σε κάποιε χώρε μέλη, στη Σουηδία α πούμε, υπάρχει νομική υποχρέωση για το κάθε σκάφο να δεχτεί τέτοιου παρατηρητέ και γίνεται κάτι τέτοιο. Ε, ανεβαίνουν οι παρατηρητέ στα σκάφη. Σε άλλε χώρε υπάρχουν άλλε προσεγγίσει. Στην Ιρλανδία, Φερρυπίν, βασίζεται αυτό σε, αυτή η συνεργασία σε, στην καλή θέληση. Αν θέλει ο καπετάνιος να τον δεχτεί τον παρατηρητή ή όχι. Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Έχουμε τα πάνω και τα κάτω μας στη συνεργασία, ανάλογα με τα θέματα. Μ' αρέσουν αυτές οι αποχρώσεις που βάζετε στην απάντησή σας. Πίτερ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχω κάποιες ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, πρώτη ερώτηση. Ο, μας είπατε ότι κοστίζουν όλα αυτά πάρα πολύ. Τι έσοδα έχει ο ISIS ανακτάτε όλα τα λεφτά τα οποία ξοδεύετε, τα οποία πληρώνετε, ας πούμε, για να ετοιμάσετε τις εκθέσεις σας. Ας πούμε, δεν κατάλαβα καλά. Ε, από αυτά που παίρνετε, ας πούμε, από την συμβουλή που, παρέγε, που παρέχετε, ας πούμε, μπορείτε να βγάλετε τα έξοδά σας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια επιστημονική επιτροπή, την STCF, Οι συμβουλές σας και η ετήσια συνεργασία σας, πώς μοιάζει, ποια είναι η σχέση σας με αυτή την επιστημονική κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την STCF. Τρίτη ερώτηση, που την άγγιξε και ο πρόεδρος Ακούω πάρα πολλά από τους ψαράδες που λένε ότι έχουν, κοιτάζουν λίγο τον Άισις και τις συμβουλές που δίνει με υποψία. Γιατί μερικές φορές θα πρέπει να προσαρμοστούν συμβουλές αυτές, παραδείγματος χάρη για τη ρέγγα της Βόρειας Θάλασσας, αλλά και άλλες και άλλα λιεύματα. Ε, και το μπακαλιάρο, ο μπακαλιάρος μειώθηκε. Γιατί λέτε ότι ε, οι ψάδε λένε πάντα έχουμε αρκετό απόθεμα. Και φυσικά είναι πρόβλημα όταν δεν γίνεται σωστή αλίευση. Οι αλίες λένε ότι πολλά από τα είδη δεν μπορούν να τα ψαρέψουν καθόλου. Βλέπουμε πολλές διαφορές με τη συμβουλή σας. Γιατί άλλα λέτε εσείς συμβουλές σας και άλλη είναι η πραγματικότητα ορισμένες φορές. Ειδικά σε ό,τι αφορά την πλατέσα. Δηλαδή, ίσως η, η ε, προσέγγιση σας από την πράξη είναι πόρο απέχει. Και δεν είσαστε κοντά στην πραγματικότητα που ζουν πολλοί αλλοίς. Για να ε, εστιάσουμε στην πλατέσα. στην κεντρική και βόρειο θάλασσα δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου πλατέσα. Επί έξι χρόνια τώρα. Βλέπω πάρα πολλές πραγματικότητες, ας πούμε, να απεικονίζονται στα όσα λέτε τελικά εσείς. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά. Βλέπουμε να υπάρχουν μια σειρά από συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θέλετε να απαντήσετε απευθείας. Ναι. Ε, ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο και η ανεξαρτησία του ΕΣΕΖ. το επιχειρηματικό μας μοντέλο της βουλευτικής συγκεκριμένα επιτροπής του ΕΣΕΖ είναι ότι τα, το κόστος το οποίο προκύπτει δηλαδή σε επίπεδο γραμματιακής υποστήριξης και ε, τους μισθούς ε, των ε, μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής που κάνουν τις διάφορες παρουσιάσεις, εξασφαλίζεται ακριβώς μέσω συμφωνιών ε, χρηματοδότησης με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ορβηγία, την Ισλανδία και ε, το, ε, οι δαπάνε των ίδιων των εμπειρογνωμόνων καταβάλλονται από τα κράτη-μέλη από τα οποία προέρχονται οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο ISIS και έχουμε μια σειρά από επιστήμονες δηλαδή οι οποίοι συμμετέχουν από διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν δηλαδή επιστήμονε οι οποίοι ε, ασχολούνται, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο απόθυμα, οπότε στι έρευνέ του εστιάζουν εκεί. Ενώ υπάρχουν ε, κάποιοι άλλε επιστήμονε οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένο ενδιαφέρον για κάποιο απόδημα και ε, απλά εξετάζουν, για παράδειγμα, κατά πόσο οι έρευνε γίνονται με βάση ε, τα ορθά επιστημονικά πρότυπα και ό,τι καθεξή. Αυτά σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό μοντέλο. Τώρα, σε σχέση με την Τεχνική και Επιστημονική Επιτροπή Αλίας τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πώ συνεργάζεται το STCF, αυτή η Επιτροπή, με το ISIS. Ε, υπάρχει καταρχήν μεγάλη επικάλυψη σε επίπεδο προσωπικού. Δηλαδή, πολλά μέλη των ομάδων εργασία του STCF είναι ταυτόχρονα και μέλη των ομάδων εργασία και των ομάδων εμπειρογνωμόνων του ΆΕΣΕΣ. Και προσπαθούμε βέβαια εδώ πολύ σκληρά να μην υπάρχει άλλη επικάλυψη των εργασιών που κάνουν η STCF και το ISIS. Στο παρελθόν υπήρξε τέτοια άλλη επικάλυψη των εργασιών μα, αλλά πρόσφατα έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ακριβώς να μην επαναλαμβάνονται ε, ίδιες εργασίες, να μην υπάρχει άλλη επικάλυψη και υπάρχει πολύ μεγάλο επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες ε, του εργασίας του STCF και τις ομάδες εμπειρογνώμων. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη μεικτή αλληλεία υπάρχει μια ομάδα του STCF που εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την διαχείριση της μεικτής αλληλείας, ενώ η ομάδα εμπειρογνωμών του αντίστοιχη του ICS ε, εξετάζει τις βιολογικές επιπτώσεις αυτών των διαφορετικών δυνατοτήτων σε ό,τι αφορά τη μεικτή αλληλεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόνοιε που έχει ο αλευτικό εκλάδο σε ό,τι αφορά τι συμβουλέ που δίνει το ISIS, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των αποθεμάτων, σε ό,τι αφορά το σκουμπρί αλλά και τη ρέγγα τη Βορειοθάλασσας Θάλασσα. πράγματι έχουν υπάρξει τέτοιου ζητήματα και εξ ορισμού ορισμένος από τι αξιολογήσει, δεν είναι αξιόπιστε. δεν υπάρχει σταθερότητα σε αυτήν την αξιολόγηση. Και το ανέφερα αυτό στην παρουσίασή μου. Δηλαδή, Εάν υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα και με συγκεκριμένα σημεία αναφορά, τότε που είναι πολύ εύκολο να γίνει μια αξιολόγηση του αποθέματο. Όμω στην περίπτωση, για παράδειγμα, του σκουμπιού, όπου έχουμε ε, κακή, α το πούμε έτσι, ποιότητα δεδομένα, για παράδειγμα, μια, μια α, α, σειρά από αναφορέ σε ό,τι αφορά τα λεμματα που ήταν ανακριβεί ακριβώ επειδή ιστορικά υπάρχει μια μεγάλη παραπληροφόρηση, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τα οποία δίνονται. Δεν είχαμε καλή αξιολόγηση τη δυναμική. Και μετά υπήρξαν κάποιε έρευνε ε, οι, οι οποίε έδειξαν διαφορετικέ διακυμάνσει σε διαφορετικέ χρονικέ περιόδου ε, και κάποιε από αυτέ ε, οδήγησαν ακριβώ σε πολύ διαφορετικέ εκτιμήσει σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αποθέματος και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τις αξιολογίες και εμείς κάνουμε μια δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, το Μάιο, για παράδειγμα, έλαβε χώρα ένα workshop σε ό,τι αφορά τον χάρτη πορεία σε επιστημονικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τι επιστημονικέ ανάγκε για την αξιολόγηση των αποθεμάτων του σκουμπριού. Και εκεί ακριβώ εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε πιο αξιόπιστε τι αξιολογήσει των αποθεμάτων σκουμπριού. Σε ό,τι αφορά τώρα την χωματίδα τη Βορειοθάλασσα στην πλατεία το τι γίνεται σε σχέση με τις σχετικές αξιολογήσεις. Βλέπουμε πως η αξιολόγηση των αποθεμάτων, η θνησιμότητα έχει μειωθεί και κατά συνέπεια το μέγεθος του αποθέματος έχει αυξηθεί. Και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει μια μετακίνηση από το νότο της Βορείου Θάλασσας ε, περισσότερο προς τα ανατολικά και στα βόρεια της Βορείου Θάλασσας. Οπότε βλέπουμε να υπάρχει μια διαφορά στην κατανομή του αποθέματος, πράγμα το οποίο βέβαια επηρεάζει τον τρόπο με το οποίο οι αλληλεί αντιλαμβάνονται την εξέλιξη του αποθέματο. Εμεί όμω εξετάζουμε την εξέλιξη του αποθέματο στο σύνολο τη Βορείου θάλασσα και προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε ε, εκτιμήσει σε ό,τι αφορά το σύνολο τη περιοχή και του αποθέματο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ε, αναξιόπιστες αξιολογήσεις και υπάρχουν και κάποια ζητήματα για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, ε, αύξηση του αποθέματος γιατί για παράδειγμα ο ρυθμός ανάπτυξης, δηλαδή το ίδιο το μέγεθος των ηχθών μειώνεται παρότι έχουμε αύξηση του αποθέματος. Οπότε εξετάζουμε και αυτό το ζήτημα ε, σε ό,τι αφορά τι εκτιμήσει που κάνουμε των αποθεμάτων χωματίδας και όλα αυτά βασίζονται από τα δεδομένα που μας παρέχει ο ίδιος ο αλληλευτικός κλάδος, δηλαδή δεδομένα του κλάδου και δειγματοληπτικά ε, προγράμματα. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλέ σχέσει εδώ με τον αλευτικό κλάδο εντό των κρατών μελών. Ε, και αύριο, για παράδειγμα, θα συναντήσω ε, τους εκπροσώπους ε, ε, του αλευτικού κλάδου στην Ιρλανδία. εκεί δηλαδή και εγώ συμμετέχω σε αυτή την αλεία και ακριβώς θα συζητήσουμε εκεί με τους εκπροσώπους του κλάδου τι ανησυχίε από την πλευρά των αλλαιών. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να εξετάσουμε ε, τις ε, πολύ διαφορετικές ε, απόψεις, τα όσα παρατηρεί ο κλάδος από την πλευρά του και το πώς αυτά διαφέρουν από τα δικά μας, τις δικές μας εκτιμήσεις, οι οποίες βασίζονται βέβαια στα επιστημονικά δεδομένα. Παρακαλώ, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε τον Ευρωγνώμονα για αυτή την παρουσίαση. Έχω μια σειρά από ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να θέσω ίσως να ξαναπάρω το λόγο, αλλά ξεκινώντα λοιπόν από τα εξή. Ε, νομίζω πως είναι πολύ ξεκάθαρο από την παρουσίαση που μας ε, κάνατε πως ε, το ISIS αποτελεί έναν επιστημονικό οργανισμό για την αλληλεία, ο οποίο συλλέγει ποσοτικά δεδομένα. Εκείνο λοιπόν που δεν βλέπουμε στην παρουσίασή σας ε, Ε, και επειδή μας είπατε ότι το ΆΣΙΣ προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες γενικότερα τη κοινωνική. και με βάση και τα ερωτήματα που θέσατε εσείς, ε, Πρόεδρε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά δεδομένα, τι υπάρχει. Για παράδειγμα, δεδομένα δηλαδή από οικολογικές οργανώσεις. και άλλους επιστημονικούς τομείς. Δεν υπάρχει κάτι, γιατί εστιάσατε πάρα πολύ στο γεγονός ότι ε, το ISIS ασχολείται με τα επιστημονικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την αλή, αλλά τι γίνεται από τον τομέα των κοινωνικών επιστημών και των αντίστοιχων ποιοτικών δεδομένων, γιατί και αυτό θα μας ε, οδηγούσε σε επίπεδο άσκησης πολιτικής. Άρα λοιπόν έχει αυτό ληφθεί υπόψη σας στο επίπεδο δηλαδή της εμπειρογνωμοσύνης ε, του ISIS. Από ότι αντιλαμβάνομαι υπάρχει και μια ομάδα εργασίας σε, σε ό,τι αφορά ακριβώς την κοινωνική διάσταση τη ε, της και θα ήθελα να ενημερώσετε λίγο εδώ την Επιτροπή μας προ το τι ακριβώς κάνει αυτή η ομάδα εργασίας του ΑΕΣΕΖ και το πώς οι εργασίες αυτής της ομάδας εργασίας θα τροφοδοτούν και θα επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων του ΑΕΣΕΖ. Όχι μόνο σε ποσοτικό επίπεδο, αλλά και σε ποιοτικό επίπεδο, δηλαδή προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στι κοινωνικέ ανάγκε. Απάντηση. Ναι, δεν ήθελα να δώσω την εντύπωση ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα ηχθείς και τα αποθέματα. Ε, πολλές από τις συμβουλές ε, τις οποίες ε, δίνουμε είναι, ε, προσπαθούμε ακριβώς να αλλάξουμε, να, να, να, φύγουμε λίγο, να απομακρυνθούμε από το υφιστάμενο μοντέλο των ε, CFP και των ποσοστώσεων και ούτω καθεξής. Και αυτό που προσπάθησα να πω στο τέλο τη παρουσίαση είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάζουμε εδώ που κάνουμε στο πλαίσιο τη οικολογική προσέγγισης η οποία ακριβώ περιλαμβάνει και την οικολογική αλλά και την κοινωνική διάσταση. Μέσα στο ISIS έχουμε τρει κύριους επιλώνες. Έχουμε καταρχήν το κέντρο των δεδομένων, μετά τον επιστημονικό πυλώνα, την επιστημονική διάσταση, όπου υπάρχει μια τεράστια ενεργή κοινότητα η οποία εξετάζει όλα τα ζήτημα των θαλάσσιων, των θαλάσσιων επιστημών όπου περιλαμβάνεται και ακριβώς η κοινωνική επιστήμη αλλά και οικονομικά ε, συστήματα και εδώ ε, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και μελλοντικά ε, στις ανάγκες σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων έτσι ώστε όταν θα τεθούν τα σχετικά ερωτήματα στο μέλλον σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις οικονομικές για παράδειγμα επιπτώσεις, τις, τις κοινωνικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές αλληλευτικές δραστηριότητε, να έχουμε εμεί την δυνατότητα σε επιστημονικό επίπεδο και του απαραίτητου εμπειρογνώμονε για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτέ τι απαντήσει. Δηλαδή, οι βασικέ έρευνε που γίνονται αυτή τη στιγμή να μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν και σε επίπεδο εφαρμοσμένων ε, πλέον, εφαρμοσμένη επιστήμη προκειμένου να δοθούν αυτέ οι απαντήσει. Δηλαδή, πρόκειται για μία από τις κύριες διαστάσεις ε, μέσα στη βασική μας στρατηγική, ότι δηλαδή θέλουμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση των συμβουλών που ε, εκπονεί η, ε, το ΆΕΣΙΣ. Να σας ακούσουμε από τους παράδοσους, κύριο Σαλόντε, έχει το λόγο. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ε, με ενθαρρύνει το γεγονός ε, ότι ο ίδιος ο κλάδος προσπαθεί εδώ να σα ε, βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν κοινά σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που έχετε στη διάθεσή σα, γιατί πράγματι υπάρχει ανάγκη να μην υπάρχουν τέτοιου είδου δεδομένα. Τώρα, αναφερθήκατε σε μια διαδικασία peer review, δηλαδή αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων και ότι υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδου αξιολογητέ από δική σα πλευρά. Ε, σε αυτή την περίπτωση, εξετάζετε και τα μοντέλα συλλογή δεδομένων σα ή μόνο τα μοντέλα υπολογισμού με βάση αυτά τα ε, δεδομένα, γιατί μα είπατε πω το ε, ε, βασικό στοιχείο για την εργασία σας είναι η καλή ποιότητα των δεδομένων που λαμβάνετε. Άρα λοιπόν, πόσο συχνά γίνεται αυτή η αξιολόγηση, επανεκτίμηση των μοντέλων συλλογής δεδομένων σας για να διασφαλίσετε την ποιότητά τους. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα. Αυτά τα ε, οριακά σημεία αναφορά που έχετε, πώς τα αντιπαραβάλλετε για παράδειγμα με εκείνα που υπάρχουν ε, για παράδειγμα στο παρελθόν, γιατί βέβαια αναφέρονται συχνά αυτά τα πολυζωνικά υποθέματα, δηλαδή που μετακινούνται από τη μία περιοχή στην άλλη. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε πόσο συχνά κάνετε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συλλογή των δεδομένων, κάνουμε αυτή την επισκόπηση Έχουμε την τύχη να έχουμε σωστό πλαίσιο συλλογής δεδομένων στην Ευρώπη, δηλαδή στο τμήμα το σχετικό έχουμε πολλούς ανθρώπους που εργάζονται εκεί και πολύ ικανούς. Το STCF λοιπόν ασχολείται με την ποιότητα των δεδομένων και εμείς στο δικό μας Συμβούλιο έχουμε διάφορες ομάδες εργασίας που ασχολούνται με την συλλογή των δεδομένων Έχουμε οργανώσει διάφορα εργαστήρια σχετικά για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων. Πάρα πολλή έρευνα δηλαδή έχει γίνει για αυτό το πεδίο της ε, συλλογής των ε, δεδομένων και της έρευνας Θέλουμε να βελτιώσουμε την ροή με την οποία μας έρχονται τα δεδομένα και τα στοιχεία από τις διάφορες χώρες για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις αξιολογήσεις μας. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, ξέρετε, τα στοιχεία μας τα έστελναν οι χώρες μέλη, δηλαδή τα εθνικά θαλάσσια ερευνητικά ιδρύματα, σε αθρηστικό με αθρεστικό τρόπο και δεν υπήρχε διαφάνεια για την ποιότητά τους. Τα στέλνουν όλα μαζί δηλαδή, συσσωρευμένα, αθρηστικά. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε τώρα περιφερειακή βάση δεδομένων και σύστημα εκτίμησης. Άρα τα στοιχεία θα έρχονται σε με πρωτογενή τρόπο από τις χώρες μέλη στο Ερευνητικό Συμβούλιο και θα δούμε τα ατομικά δείγματα και θα διαχειριζόμαστε καλύτερα τη διαδικασία. Θα έρχονται δηλαδή τα στοιχεία ανεπεξέργαστα. Νομίζω ότι είμαστε στην κίνηση στο στη κατεύθυνση. Τώρα για τα σημεία αναφορά και το benchmarking και για να αλλάξει ένα καθεστώς ή όχι. Σας απαντώ λέγοντας ότι εξαρτάται από το συγκεκριμένο απόθιαμα κάθε πόστε και κάθε πόσο συχνά γίνεται το benchmarking ο στόχος μας είναι να γίνεται τουλάχιστον μια φορά ανά 3 έως 6 χρόνια για κάθε ηχθή απόθεμα. Όταν όμως κάνουμε αυτό το benchmarking, επανεκτιμούμε και επαναξιολογούμε το σημείο αναφοράς εκείνη τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην παραγωγικότητα. Και όταν βλέπουμε τα σημεία αναφορά για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, βλέπουμε τις αλλαγές της παραγωγικότητας και το ποιος θα είναι ο αντίκτυπός τους στις προβλέψεις και εκτιμήσεις μας για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Δεν λέω ότι το κάνουμε συστηματικό τρόπο, αλλά το κάνουμε αναλόγως με το κατά κάθε πότε χρειάζεται κοιτούμε τα σημεία αναφοράς και κάνουμε την εκτίμηση για την παραγωγικότητα. Στην Ιρλανδική θάλασσα τα σημεία αναφοράς άλλαξαν πρόσφατα για το γάδο της Ιρλανδικής θάλασσας γιατί υπήρξε μεταστροφή και μεταβολή της παραγωγικότητας στην Ιρλανδική θάλασσα με βάση τη δουλειά που γίνεται ε, στο WK Irish Process. Και άρα είπαμε ότι είμαστε κάτω από το καθεστώς παραγωγικότητας, άρα τα σημεία αναφοράς για το γάδο αυτό της Ιρλανδικής θάλασσας πρέπει να αλλάξουν και το πράξαμε. Δηλαδή, μόλις καταλάβουμε τη διαδικασία και τις αλλαγές ε, στη διαδικασία, ε, τα συμπεριλαμβάνουμε αυτά στη σημεία αναφοράς και κάνουμε και εμείς τι αντίστοιχες αλλαγές. Ο Πρόεδρος, γιατί τα πράγματα μπορεί να στραβώσουν εξηγείται στην Επιτροπή. Δηλαδή, στο τελευταίους μήνες ακούσαμε για την κατάσταση στην Ισλανδία. Ο Πίτερ αναφέρθηκε στις διακοιμάνσεις σε σχέση με το καθεστώς για το σκουμπρί. Μετέχαμε κατάρρευση στη Βόρεια Θάλασσα παρόλο που έγιναν τεράστιες περικοπές στα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Αλλά και στη Βαλτική Θάλασσα ε, σε σχέση με τη Ρέγκα. Είχαμε πολύ μεγάλες διαφορές είναι Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε ότι ξαφνικά πρέπει να μειώσετε κατά 70% τα μέγιστα επιτρεπόμενα λέμματα γιατί τώρα ξύπνησαν οι επιστήμονες. Πώς έσφαλαν τόσο πολύ στο παρελθόν και ξαφνικά πρέπει να πούμε στον άνθρωπο να μειώσει κατά 70% αυτό που αλλιεύει. Θα σας απαντήσω. Ε, οι αξιολογήσεις δεν απαραίτητα η αλήθεια. Είναι μια αφαιρετική προσέγγιση της πραγματικότητας. Δηλαδή εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για να τα χρησιμοποιήσουμε ως αλήθειες στη διαχείριση. Λέμε λοιπόν για τον Μερλούκιο ότι για να αλλιεύει κανείς με μέγιστη βιώσιμη απόδοση πρέπει να αλλιεύει π.χ. 700 ε, τόνους και όχι παραπάνω. Αλλά στην αξιολόγηση του αχθιοποθέματος δεν, δεν είμαστε βέβαιοι για το συγκεκριμένο νούμερο. Οι, οι, οι ε, ε, εκφύσεως δεν μπορούν να είναι απολύτως ακριβείς. Εξαρτώνται από τα στοιχεία που βάζεις στη, μέθοδο για να θα βγάλεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Το παράδειγμα που δίνεται με το σκουμπρί είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πέρσι παρουσίασα τις συμβουλές για το σκουμπρί περίπου την ίδια εποχή. Είχαμε συμβουλεύσει 370.000 τόνους για παράδειγμα. Υπήρχε θέμα με την αξιολόγηση του αχθείου αποθέματος γιατί μία από τις πηγές των δεδομένων ήταν αυτή η οποία κατέβαζε την αξιολόγηση ενώ οι άλλες πηγές δεν συμφωνούσαν, την τραβούσε δηλαδή προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε αν αυτή η κατάσταση ισχύει, δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε, δεν είχαμε στοιχεία, έπρεπε να το μελετήσουμε. Και άρα βάλαμε ένα benchmarking για το σκουμπρί, και χρειάστηκε έξι μήνες από την αρχή μέχρι το τέλος για να δώσει αποτελέσματα και να δούμε αν σωστά και ορθά το πράξαμε. Και το Μάιο πέρσι λοιπόν βγάλαμε νέα συμβουλές και αυξήσαμε. Και είπαμε από 300 τόσο μπορείτε να πάτε σε 670.000 τόνους άνετα. Δηλαδή διπλασιάσαμε την ποσότητα που συμβουλεύαμε να αλλιευθεί. Και χθες στη Χάγη, στο Συμβούλιο για τα πελαγικά είδη, δώσαμε συμβουλές για 920.000 τόνους. Δηλαδή από 300.000 τόνους που συμβουλεύαμε και δεν επιτρέπαμε παραπάνω, λέγαμε να μην επιτρέπει παραπάνω, μέσα σε ένα δωδεκάμινο τους τριπλασιάσαμε την ποσότητα και τους είπαμε ψαρεύτε ελεύθερα ουσιαστικά. Ε, ε, υπάρχουν τέτοια ζητήματα με την αξιολόγηση. Κάποια από τα δεδομένα δηλαδή είναι διαμετρικά αντίθετα από τις διάφορες πηγές και το μοντέλο αξιολόγησης πρέπει να βρει τη χρυσή τομή, τη μέση λύση. Και ε, εν μεταξύ υπάρχουν αλλαγές και εξελίξεις ε, οι οποίες αυξάνουν την αβεβαιότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε αυτές τις αξιολογήσεις και να τις κάνουμε πιο στέρεες, αν θέλετε. Ε, δηλαδή, τα, οι, οι, διαχειριστικές και διοικητικές διαδικασίες να μπορούν να αποκρίνονται σε διαφορετικές πραγματικότητες. Μπορούμε να κάνουμε προσωμείωση διαφορετικών πραγματικότητων για το εκάστοτε ήχθη απόθεμα, και μπορούμε να δούμε κατά πόσο το διαχειριστικό σχέδιο ανταποκρίνεται σε διάφορα σενάρια. Αυτή είναι η τακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε και για το σκουμπρί και για τα άλλα ήδη. Ο κύριος Κόλμπερτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω αποκαρδιωθεί με την τελευταία απάντησή σας και Μιλούμε για επιστημονικές αξιολογήσεις που μπορεί να ασφάλουν, εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημά μου είναι διαφορετικό. Αναφερθήκατε στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά ως οργανώσεις μέλη και τη Ρωσία. Στους χάρτες που παρουσιάσατε και στις αναφορές στα νομοθετικά πλαίσια, δεν αναφερθήκατε στις χώρες αυτές. Αυτό το κάνατε για να απλουστεύσετε την παρουσίασή σας. Είτε δίνετε συμβουλές σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο μου ερώτημα. Στην παρουσίασή σας για τη θνησιμότητα είπατε ότι είναι δύο οι παράγοντες. Αλλιευτική προσπάθεια και φυσικά αίτια. Πρέπει να υπάρχει και τρίτος παράγοντας που είναι η μόλυνση και η ρήπανση. Ίσως το είπατε και εγώ έλειπα εκτός αιθούσης γιατί χρειάστηκε να λείψω για λίγο. Όμως, βλέπετε στοιχεία δεδομένα για τη ρήπανση, τη μόλυνση και τον αντίκτυπό της στη θνησιμότητα. Απάντηση. Πράγματι. Δίδουμε συμβουλές ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά για τα αποθέματα του Σολομού και της Φώκιας. Δεν είμαστε η βασική πάροχη συμβουλευτικών υπηρεσιών για το βορειοδυτικό Ατλαντικό ωκεανό. Έχουν δικά τους συμβουλευτικά σώματα, την ΑΦΚΟ και εθνικά ερευνητικά ιδρύματα έχουν διαφορετικό διαχειριστικό σύστημα. Όταν κάτι τους λείπει και κάτι δεν το ξέρουν και δεν έχουν προβλέψει μέθοδο, τότε στρέφονται προς εμάς. Όμω, Αμερικανοί επιστήμονες από τι ΗΠΑ και τον Καναδά δραστηριοποιούνται στις ομάδες εμπειρογνωμόνων και στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Τους καλούμε συχνά γιατί έχουν αμερόληπτη άποψη για το βόρειο ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό και άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η επιστημονική τους ε, συμβουλή και κατάρτιση. Τώρα για την παρακολούθηση του αντικτύπου της ε, μόλυνσης και της, ε, στη φυσική θνησιμότητα ομάδες εμπειρογνωμόνων εξετάζουν τον αντίκτυπο της μόλυσης και στα χθειοποθέματα και στις νόσους που παρουσιάζουν. Έχουμε μια επιστημονική ομάδα. Δεν περιλαμβάνεται στα μοντέλα αξιολόγησης χθειοποθέματων. Υπήρχε όμως θέμα, έχει γίνει δουλειά στη Βαλτική με τα PCB Έχουμε δώσει συμβουλές για τα επίπεδα αυτά ε, των PCB στη θάλασσα της Βαλτικής, αλλά δεν τα περιλαμβάνουμε de facto στις αξιολογήσεις μας για τη θνησιμότητα. Το ποσοστό δηλαδή του αντικτύπου οφείλεται στη μόλυση. Η μόλυση στον ωκεανό γενικά είναι τοπική πάντοτε. μπορεί να μην επηρεάσει το γενικότερο ηχθιαπόθεμα. Θα το επηρεάσει εκεί τοπικά, αλλά όχι στο σύνολο του πληθυσμού που διαβεί σε όλο τον ωκεανό ή που μετακινείται. Έχουμε περίεργες περιπτώσεις, για παράδειγμα στην Ισλανδία. Το 40% του αποθέματος της Ρέγκας πέθανε Είχαμε, γιατί πήγαν σε έναν, όλοι, όλο το εχθιαπόθεμα, ε, όλος ο πληθυσμός της Ρέγκας κατέφυγε σε ένα κόλπο που είχε πάρα πολύ χαμηλό οξυγόνο. Οπότε ξαφνικά έσκασαν δηλαδή εκεί όλα τα ψάρια και πέθαναν λόγω φυσικής, φυσικού αιτίου κατά τύχη. Ε, συμβαίνουν τέτοιου είδου ε, περίεργα πράγματα, αλλά δεν τα περιλαμβάνουμε ως πηγή θνησιμότητας, γιατί είναι κατεξαίρεση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Κόρμπετ, που σας κάλεσε να βελτιώσουμε τις μελέτες για τη μόλυνση και τις ε, ανθρωποϊδρολογικές επιπτώσεις. Ε, υπάρχουν πολλές μορφές μόλυνσης. Όπως είπατε χθες, Υπάρχουν οι αγωγοί, πούμε, πετρελαίου, φυσικού αερίου, ε, δυσκολίες που έχουν με τους βιολογικούς καθαρισμούς τα κράτη-μέλη, που πετάνε, τα λίματα όπως, ε, όπως είναι. Νομίζω ότι αυτό επηρεάζει πολύ τη θνησιμότητα των ψαριών. Και είναι ένας από τους λόγους που θα πρέπει να μελετήσουμε την ε, πηγή αυτή. Και ο συνάδελφος, λοιπόν, ε, ζήτησε να γίνουν πιο ενδελεχείς μελέτε για το θέμα αυτό της μόλυνσης. Κάτι άλλο τώρα, για τη βιομάζα. Εντάξει, επηρεάζει την, ε, τα αποθέματα. Αλλά και το σύστημα κυνηγού και θήτη, ε, θήτη και θυράματος. Αυτό μπορεί να επηρεάζει τη βιομάζα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Οι αλληλείς γκρινιάζουν ότι η μείωση κάποιων πραγμάτων ε, μειώνται κάποια είδη ψαριού, ας πούμε, γιατί πολλαπλασιάζονται τρομερά, ας πούμε, κάποια άλλα. Π.χ. ο τόνος. Ο τόνος τρώει κάποια άλλα είδη, ας πούμε, τα οποία αυτά ε, εξαφανίζονται. Η ανθρώπινη επίπτωση είναι σημαντική στο ηχθιαπόθεμα και προσπάθησα να το τονίσω ότι το ενσωματώνουμε αυτό στην Συμβουλή, κάνουμε εξο... ε... προβλέψεις πούμε ε... για τη ρέγγα και τη βιομάζα του αναπολικού αποθέματος ας πούμε που υπάρχει στο βυθό. Επίσης, στη Βόρεια Θάλασσα Έχουμε μια ομάδα που ασχολείται ε, με πολλά είδη. Και βλέπει, ας πούμε, πώς αλληλεπηρεάζονται αυτά τα είδη. Ε, και επειδή υπάρχει κυνήγι από κάποια είδη, ας πούμε, προς κάποια άλλα, ε, επηρεάζεται η θνησιμότητα. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τη δυναμική των διαφόρων ειδών και το κυνήγι που γίνεται από κάποια μεγάλα ψάρια προς μικρότερα ψάρια. Στη Βόρεια Θάλασσα, ας πούμε, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για, αυτά, για αυτούς τους σχετισμούς. Έγινε στη δεκαετία του 90 μια τεράστια προσπάθεια για να συλλέξουμε ε, πολλά δεδομένα από το στομάχι των ψαριών, ε, να δούμε τι έχουν φάει. Ε, τελείωσε όμως αυτή η προσπάθεια, δεν έχει επικαιροποιηθεί σήμερα. Χρησιμοποιούμε ακόμα πολύ παλιά δεδομένα για να ε, τροφοδοτήσουμε τα μοντέλα μας ε, και για μοντέλα που αφορούν πολλά είδη, θα πρέπει να έχεις οπωσδήποτε δεδομένα από το στομάχι των ψαριών, ούτω ώστε να έχεις σωστές παραμέτρους για τις αλληλεπιδράσεις αυτές. Είναι πρόβλημα, είναι πρόκληση μεγάλη, αλλά είναι σημαντικό το θέμα και νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε επιστημονικά. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Εγώ μιλάω Ολλανδικά. Εγώ δεν μιλάω, λέει ο Πρόεδρος. Προτιμώ. Έχω δύο ερωτήσεις, Πρόεδρε. Στην παρουσίαση ακούσαμε να μιλάτε για το οικοσύστημα. Κοιτάζετε τις επιπτώσεις ή πιθανές επιπτώσεις των ανεμομήλων, ας πούμε, στην Βόρειο Θάλασσα, τις ανεμογεννήτριες, ας πούμε. Ε, γιατί υπάρχουν σχέδια για να φτιάξουμε τεράστια πάρκα ανεμογεννητριών. Θα πρέπει να καταλάβουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα πάρκα αυτά των ανεμογεννητριών στα ηχθή αποθέματα. Μπορείτε να μας δώσετε μία απάντηση. Δεύτερον, δεύτερη ερώτηση για τις ε, αλλιευτικές μεθόδους. Το ISIS λέει οτιδήποτε όταν παρέχει συμβουλές για να κάνουμε πιο επιλεκτική αλίευση των αποθεμάτων. Να στοχεύουμε κάποια περισσότερο, κάποια λιγότερο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που έχω. Έχει γίνει δουλειά για τις ανεμογεννήτριες ε, στον ΆΙΣΙΣ και εξετάζουμε τις επιπτώσεις ε, από τον εγκατάσταση, την εγκατάστασή τους και τις επιπτώσεις των νέων μορφών βιώσιμης ενέργειας Ας πούμε έχουμε εγκαταστάσεις ε, για να εξάγουμε ενέργεια, να παράγουμε ενέργεια ας πούμε στη θάλασσα μέσα. Το να μελετήσουμε τα δεδομένα και να τα... Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τις επιπτώσεις. Έχουμε μοντέλα τα οποία μπορούμε να τρέξουμε για να δούμε ας πούμε την επίπτωση αυτή τη στιγμή. Γίνεται έρευνα λοιπόν και μπορεί να γίνει έρευνα. Τώρα πόσο καλά θα προβλέψουμε την επίπτωση αυτών των εγκαταστάσεων στα διάφορα ηχθιαποθέματα, αυτό είναι δύσκολο να το ξέρω. Πάντως είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Είναι ένα θέμα πάρε εδώ, σε δούνε και λαβήν. Θα πρέπει να κινηθούμε προφανώς προς μια βιώσιμη μορφή παραγωγής ενέργειας. Και θα πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις των ανεμογετριών στα αποθέματα, καθώς θα επεκτείνουμε το βιώσιο τρόπο παραγωγής ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τις αλλιευτικές μεθόδους και την επιλεκτική αλληλεία, αν δίνουμε συμβουλές για να βελτιώσουμε την επιλεκτικότητα των αλλιευτικών μεθόδων. Δεν το κάνουμε συνήθως. Δεν δίνουμε τέτοιε συμβουλέ για αυτό το θέμα. Μερικές φορές στι συμβουλέ μα υπογραμμίζουμε κάποια θέματα, ε, σημαντικά. Υπάρχουν τεράστια θέματα με την ε, επιλεξιμότητα και όταν υπάρχουν τα υπογραμμίζουμε. Όπως σας είπα στην αρχή και στην παρουσίαση, εμείς απαντάμε σε ερωτήματα. Αν το ερώτημά σας, ας πούμε, ήταν ας πούμε, από την Μάρε ή από οποιαδήποτε άλλη γενική διεύθυνση για την επίπτωση της ε, βελτίωσης της επιλεξιμότητας στα ήχθη αποθέματα, αν αυτό το ερώτημα ήταν διατυπωμένο έτσι θα μπορούσαν να το κοιτάξουν οι επιστήμονες και να δώσουν εύκολα συμβουλές. Αλλά εξαρτώμαστε από το ερώτημα. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν τα ψάρια τους αρέσουν οι ανεμογεννήτριες. Λέτε εκεί γύρω στις ανεμογεννήτριες να, να δημιουργούνται περιοχές ανάκτησης ε, και ανανέωσης του ηχθιαποθέματος. Α, ορισμένα ψάρια προτιμούν τις ανεμογεννήτριες. Εμείς έχουμε κάμερες στον πυθμένα της θάλασσας και μερικές φορές ε, γίνεται χαμός εκεί. Είναι κυψέλες ολόκληρες από ψάρια. Ε, είναι τελείως ε, διαφορετικό βέβαια και από πυθμένα σε πυθμένα. Ορισμένα μόνο ίδιοι όμως πάνε εκεί. Ας πούμε δεν πάει η ρέγκα, δεν πάει το σκουμπρί, δεν πάει ο γάδος. Πάνε άλλα είδη. Ε, κάθε είδος έχει τη δική του προτίμηση ως προς το ενδιατημά του. Θα ετοιμάστε και μία έκθεση για αυτό το θέμα, ελπίζω να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας του ISIS. Είναι πολύ πιο περίπλοκο το πώς λειτουργεί από το πώς νόμιζα. Έχετε, είπατε, 1.500 ε, εμπειρογνώμονες. Πολύ ωραία. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα μπορείτε να έχετε συνένεση με όλα αυτά τα δεδομένα. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Γι' αυτό ακριβώ μα δίνετε πάντα ένα εύρο, α πούμε, σε νούμερα. Αν δεν έχετε συνένεση, α πούμε, κάποιοι επιστήμονε λένε να πάμε πιο πάνω. Κάποιοι άλλοι, α πούμε, ε, συμβουλεύουν να πάμε πιο κάτω. Γι' αυτό δίνετε αυτό το εύρο ε, στην Κομισιόν όταν την συμβουλεύετε. Ή προσπαθείτε να φτάσετε σε συνένεση, α πούμε, ε, μέσω των μοντέλων. Το εύρος αυτό δεν έχει να κάνει με το αν φτάνουμε σε συνένεση ή όχι. Ε, μας, μας ζητήσαν να, να δώσουμε ένα εύρος ό,τι αφορά τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση στις συμφωνίες που έχουμε με την Κομισιόν. Τώρα, πώ φτάνουμε σε συνένεση. Το κάνουμε σε επίπεδο ομάδα εμπειρογνωμόνων μέσω συζήτηση. Κοιτάζουμε όλα τα δεδομένα, τα στοιχεία που έχουμε, κάνουμε μεγάλε συζητήσει και τελικά με συνένεση προσπαθούμε να συντάξουμε μία έκθεση τη ομάδα εργασία Μερικές φορές σε αυτές τι εκθέσεις υπάρχουν διαφορετικές προοπτικέ που αναφέρονται. Και αυτό είναι σωστό. Αλλά τελικά αυτές οι εκθέσεις των ομάδων εργασίας ε, δημιουργούνται με συμφωνία. Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα και αν ας πούμε μονομένο, ε, ή κάποιοι επιστήμονες δεν συμφωνούν, μπορούν να ετοιμάσουν και μία έκθεση μειοψηφία. της μειονότητας ας πούμε. Σε ό,τι αφορά την παροχή της συμβουλής αυτής καθ' αυτής. Μόνο οι συμβουλές που έχουν τη συνένεση δίδονται. Θα πρέπει να περάσουν αυτές τις συμβουλές, δηλαδή ενώπιον της ΕΙΚΟΜ, της Συμβουλευτικής Επιτροπής, πριν βγει αυτή η συμβουλή από εμά. Και θα πρέπει όλοι να είναι άνετα με αυτή την συμβουλή και να θεωρούν ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιστημονική συμβουλή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πέρυσι, α πούμε, είχαμε μια περίπτωση όπου δεν μπορούσαμε να φτάσουμε σε συνένεση για, κάποια, για κάνα δυο είδη. Αλλά γενικά αυτό το σύστημα λειτουργεί. Κύριος Μήμο. Θα μιλήσω ισπανικά. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και την πλήρη ενημέρωση που μας κάνατε. Πολύ πλήρη σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν κάποια είδη που είναι πιο εύκολο ας πούμε, να τα αξιολογήσουμε από κάποια άλλα. Ε, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ για τον σκουμπρί. Όταν μιλούσαμε για το σκουμπρί, ε, μιλούσαμε και για άλλα είδη που είναι σε βιώσιμη κατάσταση. Στο... Στη Βόρεια Ισπανία Σταματήσαμε να ψαρεύουμε στο 8C ένα είδος. Δεν συμφώνουσαν κάποιοι, κάποιοι λέγανε ότι σε καλή κατάσταση, κάποιοι όχι. Στις εκθέσεις που βάζετε που στέλνετε στην Κομισιόν για να ε, καθορίσουμε τις ετήσιες ποσοστώσεις. Αυτές οι εκθέσεις είναι όλες δημόσιες. Υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι πιο εμπιστευτικές. Ε, υπήρχε μεγάλη διαφωνία για το θέμα της καραβίδας στη Βόρεια Ισπανία. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν σε καλή κατάσταση, κάποιοι όχι. Κάποια ε, αποθέματα είναι πάρα πολύ ε, πιο εύκολο να αξιολογήσουν, κάποια πιο δύσκολο. Ας πούμε, ε, με το σκουμπρί ε, είναι πολύ μεταναστευτικό το είδος αυτό και είχαμε μεγάλες αλλαγές. Το 2010, ας πούμε, στην θάλασσα της Νορβηγίας, ε, βρισκόταν εκεί, μετά την, το 2010 πήγε πιο δυτικά στα ύδατα της Ισλανδίας και της Γρυλανδίας και ίσως και πιο πέρα. Αυτές οι μεταναστεύσεις δεν είναι σταθερές στον χρόνο, διακυμαίνονται. Πέρυσι τα ψάρια αυτά επανήλθαν στη θάλασσα της Νορβηγίας. Και επομένω είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε ας πούμε, την ε, κατάσταση αυτού του συγκεκριμένου είδους, γιατί μετακινείται πάρα πολύ γρήγορα. Για ένα πελαγικό είδο. Ε, έχουμε ακουστικές έρευνες για να μελετήσουμε την βιομάζα του αποθέματος. Γιατί όταν ε, μετακινείται τόσο γρήγορα, δεν μπορείς να το πιάσει τη σωστή στιγμή, ούτως ώστε να κάνεις την ακουστική μελέτη, ας πούμε, τη σωστή χρονική στιγμή. Υπάρχουν διάφορε έρευνε που γίνονται. Γενικά τα αποθέματα έχουν, που έχουν μεγάλε ανανεώσεις στον πληθυσμό έχουν συγκεκριμένα γεωγραφικά πεδία ε, και τότε είναι πιο εύκολο να τα αξιολογήσουμε γιατί έχουμε καλά στοιχεία στα δεδομένα και δεν υπάρχει μετανάστευση εύκολα. Δεν φεύγει το είδος από το συγκεκριμένο μέρος, δεν έρχονται νέα δεν γίνεται ανανέωση του πληθυσμού, σε ό,τι αφορά ε, την Καραβίδα στη Γαλλικία, στη Βόρεια Ισπανία δηλαδή, εκεί το, το απόθεμα έχει μειωθεί ο πληθυσμό του συντο χρόνο. Ο, εν μέρη λόγω αλίας, εν μέρη λόγω περιβαλλοντικών αιτιών. Δηλαδή έχουμε αδύναμη ανανέωση του πληθυσμού ε, επί χρόνο. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε υποθαλάσσια ε, επισκόπηση, λήψη, για να έχουμε καλές εικόνες για την πυκνότητα του αποθέματος και από ό,τι φαίνεται λειτουργεί πάρα πολύ καλά ε, στην Ιρλανδία, στη Σκοτία, στα είδατε αυτά και αλλού στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή η μέθοδος δηλαδή. έχουμε μια επιλογή από εργαλεία για να αξιολογήσουμε το απόθεμα. Δεν έχουμε τέτοιε πληροφορίε και τέτοια είδη δεν χρησιμοποιούμε ακόμα στη Βόρεια Ισπανία. Επομένω, δεν έχουμε ακριβή ιδέα για το τι συμβαίνει με το είδος αυτό, με την καραβίδα αυτή, ε, υπάρχει ένα σχέδιο ανάκτησης και μηδενική, μηδενική, μηδενικό τάκ επί χρόνια. Ε, δεν έχουμε και πολλές πληροφορίες και από τη δειγματοληψία από το είδος αυτό. Έχουμε λίγες πληροφορίες λοιπόν για να αξιολογήσουμε, για να δούμε αν υπάρχει ανανέωση του, και ανάκαμψη του είδους αυτού, του αποθέματος αυτού. Επομένω, χρειάζονται περισσότερα δεδομένα και περισσότερη δουλειά για αυτό το απόθεμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει, ποια είναι η δυναμική του, ποια είναι η κατάστασή, σου, η κατάστασή του. Αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα έτσι πολύ μεγάλα όπως αυτό με το σκουμπρί, αλλά γενικά εξολογήσεις σας βελτιώνονται, ρωτάει ο Πρόεδρος. Απάντηση. Ναι, θεωρώ πως οι αξιολογήσεις μας βελτιώνονται με την ε, πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν δηλαδή μέθοδοι ούτως ώστε οι εκτιμήσεις μας ε, να γίνονται και πιο διαφανείς και λέξιμες. Και εδώ επαναρχόμαι και στο τελευταίο ερώτημα που τέθηκε. Ω προ το κατά πόσο δημοσιεύονται τα πάντα. Ναι, όλε οι εκθέσει των ε, ομάδων εργασία δημοσιεύονται. Μιλάμε για πολύ μακροσκελείς εκθέσεις, πολύ τεχνικές, αλλά είναι όλες τους διαθέσιμε δημοσίως και ίσω υπάρχει και σωρία, υπερβολική σωρία πληροφοριών από την πλευρά του ΆΣΕΣ, γιατί πραγματικά μπορεί κανεί να βρει εκεί πράγματα τα οποία δεν ήξερε ότι υπάρχουν. Υπάρχουν μία σειρά από πολύ χρήσιμα έγγραφα λοιπόν. Όλες, ε, όλα λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μα ε, και όλε οι αξιολογήσει δημοσιεύονται και είναι δημοσίω διαθέσιμα όλα αυτά. Ε, και εργαζόμαστε και ε, μέσα σε ένα πλαίσιο ε, διαφάνειας. Δηλαδή όλα τα δεδομένα που τροφοδοτούν τις εκτιμήσεις αλλά και τα output data, δηλαδή τα συμπεράσματα που βιώνουμε από αυτές τις εκτιμήσεις είναι όλα τους δημοσιευμένα. Οπότε θεωρώ πως το ΆΣΙΣ πραγματικά είναι μια πάρα πολύ διαφανής οργάνωση. Είναι η κυρία η τελευταία μιλήτρια που έχω. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Εγώ τέσσερα σημεία θα ήθελα να δείξω. Καταρχήν, ε, θεωρείται πως ένας μεγαλύτερος ε, ε, στόλος από μικρότερα αλληλευτικά σκάφη, δηλαδή λιγότερο από 10 και 15 μέτρα, είναι καλύτερα για την διατήρηση των αποθεμάτων και των οικοσυστημάτων, σε αντίθεση με τα πολύ μεγάλα αλληλευτικά σκάφη, όπως για παράδειγμα τα πολύ μεγάλα αλλιευτικά σκάφη που αλλιεύουν αυτή την περίοδο από τον κόλπο του White. Επίσης, υπάρχουν κάποια αποθέματα τα οποία βρίσκονται σε, σε μείωση. Μάλλον δηλαδή πρόκειται για κακή πρακτική από την πλευρά των τοπικών αλλιέων, με βάση δηλαδή τα λανθασμένα εργαλεία. Από εκεί και μετά τρίτο ερώτημα. Σε ό,τι αφορά ε, την, ε, τα αποτυχημένα αποτελέσματα της ε, έρευνας σε ό,τι αφορά την άκρα και τα δεδομένα που βασίζονται στα δεδομένα των τοπικών αλλιέων. θα ήθελα να ρωτήσω, αφού λέμε ότι γενικά δεν πρόκειται για αυτό μόνο που αλλιεύουμε και για τα όσα θανατώνουμε, πώ πώς αξιολογούνται γενικότερα εθνισμότητα και άλλων ειδών ε, σε αυτά τα οικοσυστήματα. Επίσης, υπάρχει περιβαλλοντικό, περιβαλλοντική βλάβη που προκαλείται από, τα από τον αλευτικό ε, στόλο, γιατί οι σχετικέ ποσοστώσει είναι υπερβολικές και επειδή τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα θέτουν σε κίνδυνο ε, είδη τα οποία ήδη απειλούνται από εξαφάνιση, που είναι ήδη απειλούμενα. Παρακαλώ. Ο κύριος ε, Λόρνταν θα πάρει το λόγο, ναι. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, θα προσπαθήσω να το αποφύγω. Εντάξει, ε, το ερώτημα που θέσατε, θέλουμε πολλά μικρά αλλιευτικά σκάφη, ε, λιγότερα αλλά μεγαλύτερα αλλιευτικά σκάφη. Δεν είναι αμυγός επιστημονικό αυτό το ζήτημα, δεν έχω πραγματικά μία θέση από αυτού. Εμείς δίνουμε συμβουλές σε ό,τι αφορά το γενικότερο επίπεδο θνησιμότητας, ε, με βάση δηλαδή και την αλληλευτική προσπάθεια. Αυτό αξιολογούμε εμείς δηλαδή. Το πόσο, πώς θα γίνεται αλληλεία, δηλαδή σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα για παράδειγμα των συγκεκριμένων ειδών που αλεύονται και το είδος του στόλου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τις διάφορες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του, της σύνθεσης του στόλου. Δεν μπορούμε δηλαδή να δώσουμε συμβούλες από πλευρά του ΆΕΣΕΣ από αυτού. Δηλαδή, ε, ανάλογα με τα διαφορετικά καθεστώτα αλίας που υπάρχουν σε διαφορετικές περιοχές ε, ε, του κόσμου, χρησιμοποιούνται ή μικρότερου μεγέθους αλευτικά σκάφη, μεγαλύτερου στο στόλο, εξαρτάται δηλαδή από την κάθε περιοχή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα αρκετά μεγάλο στόλο και προσπαθούμε κάπως να τον εξορθολογήσουμε εδώ και σειρά ετών και ίσως έχει περισσότερο νόημα να εξορθολογήσουμε λοιπόν αυτόν τον στόλο με την έννοια του ότι από τη μία πλευρά με μικρότερα αλλιευτικά σκάφη έχουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης αλλά κάποια για πελαγικά είδη όπως για παράδειγμα ε, το σαβρίδι ή το σκουμπρί ή η ρέγγα η Ρέγκα ε, αλλιευονται από, και καλύτερα και αποτελεσματικότερα από μεγαλύτερου μεγέθους αλλιευτικά σκάφη. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του λαβράκιου. Ε, πρόσφατα στην Βόρειο Θάλασσα, κανάλι της Μάχης, ε, ανατολική ε, θάλασσα της Ιρλανδίας. Εκεί λοιπόν οι αξιολογήσεις έδειξαν ε, μια περίοδο πολύ χαμηλών επίπεδων ανανέωσης του αποθέματος. Βλέπουμε τώρα πολύ πρόσφατα μια, κάποια ανάκαμψη της ανανέωσης και ανταπόκριση σε αυτή την ανανέωση του αποθέματος και εμείς από πλευρά του Άισες, λοιπόν προτείναμε μια πολύ σημαντική μείωση του αλληλήματος κατά τα τελευταία δύο χρόνια και πρόκειται για μια αξιολόγηση η οποία έχει ε, δει και κάποιες διακυμάνσει, δηλαδή σε κάποια έτη προτείναμε μηδενική αλία και σε κάποια, άλλη, ε, κάποια άλλα έτη επιτρέψαμε με κάποια αλία, δηλαδή οριακά βρισκόμαστε εκεί και δεν ήταν πραγματικά πολύ σταθερή η αξιολόγηση που παρήχαμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση βλέπουμε κάποια σημάδα, σημάδια ανάκαμψης ε, του αποθέματος αλλά ειδικότερα η Επιτροπή και άλλοι έχουν ε, προτείνει να μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό τη στοχευμένη αλεία του λαβραδιού, ειδικότερα ε, και στο επίπεδο και τη ερασιτεχνική αλεία να υπάρξουν ε, περιορισμοί. Και συμφωνώ σίγουρα με αυτό που είπατε, ότι δεν, έχει, δεν παίζει ρόλο ακριβώ το τι αλεύουμε, αλλά και το τι θανατώνουμε τελικά, δηλαδή το τι εκφορτώνουμε ω αλεύμα και τα παρεμπίπτοντα. Και εμεί κάνουμε από την πλευρά μα ό,τι μπορούμε ώστε να ε, μετρούμε και τα απορριπτόμενα αλλιεύματα μαζί με τα παρεμπιπτόντα. Γιατί παρότι απαγορεύεται ήδη η απόρριψη, παρόλα αυτά λαμβάνει σε κάποιο βαθμό απόρριψη αλλιευμάτων ε, στα χωρικά δεδομένα της Ένωσης. Και προσπαθούμε, όπως είπα ήδη, να εξετάζουμε τις γενικότερες επιπτώσεις ε, των αλλιευτικής δραστηριότητας ε, στα θαλάσσια, στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα οικοσυστήματα για να βλέπουμε ποιες είναι οι σωρευτικές επιπτώσεις δηλαδή της αλληλείας στα αποθέματα αλλά και στο ευρύτερο βιολογικό θαλάσσιο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Δύο συντονιστές μόλις προσήλθαν εδώ. Η κυρία Σάλεβεν νομίζω πως θέλει να δευτερολογήσει. Γνωρίζουμε βέβαια όλοι μας ότι ο κύριος Λόρνταν εδώ αγορεύει και παντές ερωτήματα εδώ και δύο ώρες. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέει κυρία Σάλεβαν, ε, σας ευχαριστώ που αναφέρατε ήδη και εσείς ότι θα είμαι σύντομη. σε ό,τι αφορά το ανώτατο όριο, το ανώτερο όριο του σημαίνει αναφορά για, το, για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αλλά για το 2019 για τη Ρέγκα, το ΤΑΚ τέθηκε ακριβώς με βάση το ανώτερο MSY. Για τον ε, Μερλούκιο λοιπόν δεν ε, υπάρχει μια τέτοια πρόθεση να προταθεί δηλαδή με βάση το ανώτερο MSY. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Θεωρείτε πως κάτι τέτοιο είναι βιώσιμο. Και δεύτερον, ε, η αλία της Ρέγκας έχει απαγορευτεί από το Υπουργείο της Ιλλανδίας στην, στην τη της Ιλλανδίας, αλλά αυτό έγινε πολύ αργά, η απαγόρευση δηλαδή. Ποια είναι η άποψη του σε ό,τι αφορά τα αποθέματα ρέγκα εκεί. Στα πολιετή σχέδια αλίας έχουμε προβλέψει αυτά τα περιθώρια έτσι ώστε να υπάρξουν ε, δηλαδή αυτές τις αυσομοιώσεις ό,τι αφορά την ε, μεικτή αλία και την αλία διαφορετικών ειδών, πολλαπλών ειδών. Ε, σε ό,τι αφορά το ανώτερο, όπως είπαμε, σημείο αναφοράς του MSY, θεωρούμε πως είναι έχει και την προληπτική προσέγγιση με βάση τις δικές μας ε, προσωμιώσεις, αλλά δεν θα προτείναμε να χρησιμοποιηθεί ε, αυτό το ανώτερο σημείο του MSY για όλα τα αποθέματα. Όχι, αυτό, ε, δηλαδή το σκεπτικό είναι ότι αξιοποιεί κανείς αυτό το, το σημείο εφόσον υπάρχει μία, ένας περιορισμός σε ό,τι αφορά το ΤΑΚ με μία αυξομοίωση εκεί της τάξης του 20%, περισσότερο ή λιγότερο 20%. σε ό,τι αφορά τώρα και τις επιπτώσεις σε άλλα είδη, δηλαδή εάν υπάρξει αυξημένη θνησιμότητα η οποία μπορεί να επηρεάζεται και από τον ανταγωνισμό μεταξύ των ειδών, ενδεχομένως να έχει νόημα για ένα συγκεκριμένο απόθεμα να μειωθεί σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Και βέβαια στην, ε, στην ε, πολλαπλών ειδών υπάρχει και ο στόχο ακριβώ του να μειώνονται τα παρεμπίπτωτα αλλιεύματα. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα περισσότερα που είπαμε και συγκριτικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω ότι υπήρξε μια τέτοια συμβουλή σε ό,τι αφορά την ε, ρέγγα τη ε, Βαλτική, ότι δηλαδή να αξιοποιηθεί αυτό το ανώτερο ε, MSY. Πάντω ε, στο παρελθόν έχει ζητηθεί από το ISIS να γνωμοδοτήσει επί του κατά πόσο, ειδικότερα στην περίπτωση της Βαλτικής αυτή η θάλασσα που στοχεύει πολλαπλά ήδη θα δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη το ανώτερο MSY. Πέρσι λοιπόν η δική μας άποψη ήταν ότι δεν υπήρχε κάποια ένδειξη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αυτό το απόθεμα το ανώτερο MSY. Οπότε υπάρχει συμβουλή που δίδεται από, την, από το ISS. Σε ό,τι αφορά τώρα ευρύτερα περιθώρια, μπορεί κάτι τέτοιο να ε, επιτρέπεται σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα αποθέματα και από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά η Ρέγκα στην, ε, στην θάλασσα της Ιλλανδίας Υπάρχει ακόμα κάποια ποσότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί για το 2019. Νομίζω πως η απαγόρευση στην οποία προέβη το Υπουργείο της Ιλλανδίας ε, ήταν πολύ σωστή. Και από την πλευρά δηλαδή του κλάδου να θέλει να περιορίσει σημαντικά την αλία για το 2019 αφού βλέπουμε να υπάρχουν και κάποια σημάδια αυξημένη ανανέωση του αποθέματο. δηλαδή η περίοδος αλλιώς ξεκίνησε πριν από δύο, τρεις εβδομάδες και είδαμε να υπάρχει μεγάλη αλίευση των ηχθείων κάτω από 20 ε, εκατοστά που σημαίνει ακριβώς ηχθίδια νέα ε, ε, ψάρια. Πράγμα βέβαια το οποίο καταδεικνύει ότι υπάρχει ακριβώ μια θετική εξέλιξη, δηλαδή υπάρχει μια ανανέωση του αποθέματος. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λόρντεν. Έχουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ε, είστε υποχρεωμένοι να μιλήσετε, αλλά αν επιθυμείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο, παρακαλώ έχετε το λόγο. Μόνο αν ε, θέλετε κάτι να πείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλουμε να ενημερώσουμε την Επιτροπή για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Παίρνουμε απλά το λόγο για να πούμε ότι η παρουσίαση ήταν εύγλωτη από μόνη της δείχνει πόσο στέρεα πρέπει να είναι η εμπειρογνωμοσύνη για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αξιολογήσεις. Δείχνει το πόσο μεγάλη δουλειά και πολλή δουλειά γίνεται στο Ερευνητικό Συμβούλιο το Διεθνές για την εξερεύνηση της θάλασσας και πόσο περίπλοκα είναι όλα αυτά. Πόσο περίπλοκη είναι η αξιολόγηση των επιστημονικών πορισμάτων και η διαχείριση της κατάστασης επιτόπου αλλά και η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων. Σε κάθε περίπτωση είναι απολύτω απαραίτητο να συνεχίσουμε να συλλέγουμε στοιχεία και δεδομένα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο σε Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λόρνταν που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας και που μας δώσετε τόσο συνολικές απαντήσεις μου εμπεριστατωμένα. Σας παρακαλούμε να μην μας φέρνετε ε, επιστημονικές συμβουλές με πάρα πολύ ευρύ φάσμα, γιατί ως πολιτικοί δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε μία τιμή. Ελπίζω να, να συνεχίσετε να έχετε θερμές σχέσεις με τους αλλοίς ανά την Ευρώπη. Λοιπόν, Προχωρούμε στο έργο μας. Έχουμε τον κατάλογο των προτινόμενων εκθέσεων ίδια πρωτοβουλίας και έχει γίνει μια κάποια παρανόηση εκεί. Νομίζω ότι εδώ είναι όλοι συντονιστές και μπορούμε αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είχα καταλάβει ότι είχαμε συμφωνήσει ότι η πρόταση του ΕΛΚ για τα αιωλικά πάρκα θα μπει στο 6. Θα κρατήσουμε τις δύο εκθέσεις για την απασχόληση. Τη μία, όπως είπε και ο κύριος Φερέιρα, τη μία για τις παράκτιες κοινότητες και την άλλη για την απασχόληση στα ελευτικά σκάφη και θα βάλουμε την πρόταση της κυρίας Κόντε για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση ως πρώτη εναλλακτική. Έτσι είχα καταλάβει εγώ. Κάποιοι άλλοι εσείς το έχετε καταλάβει διαφορετικά. Να δώσω το λόγο στην κυρία Κόντε καταρχάς. Υπάρχει ένα mail που ζητάει να μπει η πρότασή μου ε, στον κατάλογο μαζί με την πρόταση Φερέιρα. Στα πλαίσια ενός συμβιβασμού ε, δέχεται να αποσύρει την πρότασή του και να τη βάλει στο pipeline και να βάλει τη δική μου αντί της δικής του. Ε, με δύο λόγια δηλαδή, να αντικαταστήσει τη δική μου πρόταση, ε, με τη δική μου πρόταση την πρόταση Φερέιρα. Να μπει η δική μου πρόταση αντί για την πρόταση Φερέιρα, στο νούμερο, στο νούμερο 4. Αν συμφωνεί ο κύριο Φερέιρα, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Um, Οι άλλοι συντονιστέ είναι ικανοποιημένοι με αυτή την πρόταση. Στον κατάλογο Περιλαμβάνονται τα ολικά πάρκα του ΕΛΚ, λοιπόν, για τις έξι εκθέσεις ίδιες πρωτοβουλίας, το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, να μου το επιβεβαιώσετε. Λοιπόν, Μαύρη Θάλασσα πρώτον. Δεύτερον, αντίκτυπο των νεολικών πάρκων που είναι στην ανοιχτή θάλασσα. Μετά, ε, τα, η ρήπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον και τα σκουπίδια. Μετά, το θέμα των αλλιευτικών κοινοτήτων και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει την τοπική και αλληλεία και πώς θα αναπτύξουμε περισσότερες περιοχές για την ανανέωση των αποθεμάτων σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές, ούτως ώστε να λειτουργήσουν ως ζώνες οτοκίας και οφορίας. Ε, πρόταση δηλαδή τώρα είναι της κυρίας Κόντε για την άνοδο της θερμοκρασίας της στάθμης των ωκεανών και τη συνέπειες, στα, το αντίκτυπο στα αποθέματα θα περιληφθεί, θα συμπεριληφθεί αυτό και υπάρχει πρόταση έκθεσης για προσέλκυση των νέων για να στελεχώσουν τα αλληλευτικά σκάφη και να δημιουργηθεί απασχόληση για τις αλληλευτικές κοινότητες. Δεν είναι έτσι, κυρία Αγγιλέρα, παρακαλώ. Όχι. Αυτό που είπατε για την απασχόληση είναι δική μας πρόταση των σοσιαλιστών. Αν θέλει κάτι να αποσύρει ο κύριος Φαϊρέιρα, να αποσύρει το δικό του, όχι το δικό μας.

We have, we are having, have... Λοιπόν, ίσως υπήρξε πρόβλημα με τη μετάφραση ή την ερμηνεία, δεν είμαι σίγουρος, λέει ο πρόεδρος. Κυρία Κόντε, μας τα ξαναλέτε παρακαλώ. Εγώ έκανα λάθος. Είναι η παριθμόν 25 η πρόταση του κυρίου Φερέιρα. So, you... 4. Είπα 4, αντί για 25. Καλώς. Άρα, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, προσελκύουμε τη νέα γενιά στελεχών στο δαλευτικό σκάφος και δημιουργούμε θέση απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες. Αυτό παραμένει και είναι δικό σας, κυρία Αγγιλέρα, και είναι και το τελευταίο. Καλώς. Όχι, το τελευταίο είναι πώς θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, την ερασιτεχνική και τοπική αλληλεία. Αυτό θα πάει ως πρώτο αναπληρωματικό στην, στην αναμονή και την έκτη και τελευταία θέση θα καταλάβει η πρότασή σα για την άνοδο της θερμοκρασίας στη... της στάθμης και το καθεξής. Ο κύριος Κάλσκιν. Συμφωνώ. Όμως, στα... στις αναπληρωματικές εκθέσεις υπάρχουν και άλλα θέματα. Άρα, αν βάλουμε την πρόταση στην πρώτη σειρά, τότε θα ήθελα να εγκρίνουμε τις δύο επόμενες. Πρόταση του Ρινιού. Τη κατάσταση για την εφαρμογή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και τις υπόλοιπε οπτικές. Τότε θέλω να εγκρίνεται ότι είναι δεύτερη αναπληρωματική έκθεση αυτή για την κοινή αλληλευτική πολιτική στη δεύτερη θέση να τον εγκρίνετε και να την κατακυρώσετε για να δεχτώ να μπει στην πρώτη θέση των απληρωματικών η έκθεση της κυρίας Κόντε. Κοιτάξτε, πάντοτε έχουμε καταλόγους αναπληρωματικών, αλλά δεν είχαμε προτεραιότητες, δεν ήταν με λίστα αρρύθμισης. Οι συντονιστές, όταν υπάρχει χώρος, αποφασίζουν ποια από τις αναπληρωματικές θα μπει και θα εγκριθεί. Δεν έχουμε δηλαδή αριθμητικό κατάλογο σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση στα αναπληρωματικά. Προτείνω το, η έκθεση του κ. Φεραίρα να πάει στι αναπληρωματικέ χωρί αριθμό, ούτε η δική σα. Ο κ. Ναι, αλλά δεν είπατε αυτό. Είπατε ότι την έκθεση αυτή τη βάζουμε στην πρώτη θέση των αναπληρωματικών. Και αν λέτε πρώτη θέση στι αναπληρωματικέ εκθέσει, σημαίνει ότι υπάρχει δεύτερη. Άρα ή θα πείτε ότι θα μπει στο κατάλογο ε, των αναπληρωματικών και τέλος ή θα μπει στην πρώτη θέση. Και αν μπει στην πρώτη θέση, τότε εγώ επιμένω η άλλη έκθεση για την κοινή ελευτική πολιτική να μπει στη δεύτερη θέση. Να είστε ακριβείς. Κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρο, μου ασκεί κριτική και ο συντονιστή από τη δική μου ομάδα και προσπαθώ να λειτουργήσω με διαφάνεια. Ό,τι και να πω για πρώτη και δεύτερη θέση, τότε μιλούμε για ένα κατάλογο ενδυνάμει εκθέσεων που μπορούν να εξεταστούν ότι σε έφθετο χρόνο εάν χρειαστεί κάποια να γίνει και υπάρχει χώρος για να γίνει. Ικανοποιήστε με την εντυμότητά μου, τουλάχιστον με την ειλικρίνεια εννοώ. Ευχαριστώ. Άρα, να υιοθετήσουμε τις συστάσεις των συντονιστών. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, μπορούμε να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ τη συνεδρίαση. Να σας πω ότι στις 12 Νοεμβρίου θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ πρόεδρος τότε. Και αν δεν είμαι, θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς και τη γραμματεία. Ευχαριστούμε και εμείς για όλη αυτή τη βοήθεια που μας έχουν δώσει. Ευχαριστώ τους αντιπρόεδρους και τους συντονιστές για τη δουλειά τους. Ευχαριστώ όλους.